Συνάδελφοι, αρχίζουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Πάμε. στην ε, θέσπιση ενός ε, οργάνου για την ε, σταθερότητα. Η Φρανσίσκα Καταρίνα Μπράντνερ είναι η συγγήτρια. Μία ώρα περίπου θα κρατήσει η συζήτηση, θα τελειώνουμε μέσα σε αυτή την ώρα και είναι μία συζήτηση που θέλει να προετοιμάσει το σχέδιο έκθεσης για το σχέδιο σταθερότητας που θα συζητηθεί στις 30-31 Μαΐου στην ΑΦΕΤ. Είναι το μόνο πρόγραμμα που έχει στη διάθεσή της η Ένωση για να απαντήσει στις ε, κρίσεις και στα προβλήματα ασφάλειας ε, σε περιφερειακό επίπεδο θέλει να κάνει, να, να, σταθ, παλέψει για το, την οικοδόμηση της ειρήνης, για την σταθερότητα και για τη διατήρηση της ασφάλειας. Λοιπόν, να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και μετά την εισηγήτρια. Τέσσερα λεπτά ο κάθε εμπειρογνώμων, η δόκτωρ Μαρτινέλη, ο κύριος Σέριφ, ο κύριος Μπεν Μουρ, και η κυρία Ροζάνα Κριστέσκου. Η Δόκτωρ Μαρτινέλη από το Open Society Institute. Καλό απόγευμα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να λάβω το λόγο σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για το μέσο σταθερότητος. Μου ζητήθηκε να εστιάσω στα ισχυρά και τα αρνητικά σημεία αυτού του μέσου. Βέβαια γνωρίζουμε ήδη τα αρνητικά σημεία, το ότι το εργαλείο αυτό δεν έχει γεωγραφική δέσμευση, δεν δεσμεύεται με κριτήρια για την οργάνωση που αφορά τη δημοκρατία, εστιάζεται σε αιστείες κινδύνου και αντιμετωπίζει την ε, πρόληψη συγκρούσεων. Θέλω να αναφέρω καταρχήν ορισμένα θέματα σε σχέση με την ανάληψη κινδύνων. Υπάρχει ένα γενέ στοιχείο ανάληψη κινδύνου το οποίο δεν αναπτύσσεται πλήρω στην πρόταση αυτή. 70% των κονδυλίων θα χρησιμοποιηθούν για συνεχιζόμενες ή αναδυόμενες κρίσεις. Και κατά την άποψή μου, η διαβούλευση με τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, <clears throat> βρίσκονται, βρίσκονται σε επίπεδο ελλειπές. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν σε μια τοπική συμμετοχή των ε, εμπλεκομένων σε μεγαλύτερο βαθμό ώστε να μειώσουμε τους κινδύνους αλλά να είμαστε και έτοιμοι για το γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχει τοπική συμμετοχή και να προκύψουν ως ε, εξ αυτού προβλήματα και επίσης να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ε, πληροφόρησης και παροχής εκθέσεων για τα θέματα αυτά. Ένα δεύτερο σημείο είναι η καλύτερη συνεργασία των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αντιπροσωπιών της Υπηρεσίε Εξωτερική Δράση και των εργαλείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τι δυνατότητε που μα δίνει η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, <clears throat> ιδίω σε ό,τι αφορά τι σχέσει τη με τι οικονομικέ υπηρεσίε σε επίπεδο κεντρικού αρχηγείου, αλλά επίση και μεταξύ τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και των επιτοπίων αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν οι αντιπροσωπείε λοιπόν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην πρόταση αυτό, αυτή. Έχουν μια καλύτερη σχέση για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ιδίω όταν μπορούν να δώσουν έγκαιρη και συνεκτική πληροφορία για τις επιτόπιες συνθήκες, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία προτεραιοτήτων και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την κατανομή πόρων. Επίσης για την παρακολούθηση οι αντιπροσωπείες μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν στοιχεία για τις επιτόπιες δαπάνες και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν αναλυφθεί. Τρίτο σημείο που θέλω να δείξω. <clears throat> Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και εκθέσεις. Γενικά θεωρείται ότι είναι επιτυχές αυτό το εγχείρημα και ορθά. Πρέπει να σκεφτούμε όμως περισσότερο για το να αναπτύξουμε περαιτέρω την αξιολόγηση, όχι μονάχα σε επίπεδο κονδυλίων και βαθμού εκτέλεσης, αλλά να φτάσουμε και στα πραγματικά αποτελέσματα που επιτυχάνουν τα σχέδια τα οποία υποστηρίζονται από το πλαίσιο αυτό. Παραδείγματο χάρη, ποιο είναι ο τρόπο με τον οποίο τα προγράμματά μα ανταποκρίνονται σε επιτόπιε αλλαγέ και πώ μπορούμε να δείξουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία από την άποψη αυτή. Να αναφέρω ιδιαίτερα τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύω ότι η αξιολόγηση από εξωτερικούς συμβούλους δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει και η κοινωνία των πολιτών να εμπλέκεται περισσότερο με διαβουλεύσεις για την παροχή εκθέσεων και θα πρέπει να συμβάλλει στις εκθέσεις αυτές. Δεν ξέρουμε ακόμα με ποιο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη μνήα για την κοινωνική συμμετοχή. Θα μπορούσαν λοιπόν να είναι τμήμα της διαδικασίας διαβούλευσης και αξιολόγησης και να αρρωγούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης προβλέπεται στο σύστημα αυτό μια εταιρική σχέση για την οικοδόμηση της ειρήνης. Αυτό λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συστηματοποιηθεί περισσότερο η συμμετοχή του IFS. Επιπλέον, στο παρελθόν το μέσο αυτό δεν έχει κάνει ίσω την καλύτερη χρήση των διεθνών φορέων για να υποστηρίξουν την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να αποθαρρυνθεί η χρήση υπεργολαβιών όσο είναι δυνατόν και να υπάρξει μια πιο άμεση σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Τέταρτο και τελικό σημείο, σχέση μεταξύ μέτρων κατά της τρομοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εμπειρία του Ιδρύματός μας σε διαφορετικές χώρες στο κέρας της Αφρικής δείχνουν ότι αυτά τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας δημιουργούν έφορο έδαφος για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειώνουν τη δυνατότητα δράσης των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ένας από τους ε, στόχους του μέσου αυτού είναι να προωθήσει την αντιτρομοκρατική νομοθεσία και εδώ θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να παίξει κάποιο ρόλο ως διαμεσολαβητής μεταξύ της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και έτσι θα ήθελα να τονίσω ότι σήμερα υπάρχει ένας στεναρός μηχανισμός παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Yes, um, thank you very much. Um, Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Θα σας παρουσιάσω κάποιες μελέτες ε, στις οποίες συμμετείχα, εξετάζοντας ε, το, το μέσο σταθερότητα και πώς διαμορφώνεται σε πολλές χώρες. Νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να πούμε για το μέσο σταθερότητα είναι ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο για την πρόληψη συγκρούσεων, ωστόσο δεν είναι το μόνο. Και υπό την έννοια αυτή είναι σημαντικό η οικοδόμηση της ειρήνης και η αποτροπή συγκρούσεων να μην στερηθεί τα υπόλοιπα μέσα τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν από το DCI και το Ευρωπαϊκό Μέτρο Γυπνίασης, Μέσο Γυπνίασης. Γιατί αν θέλουμε μακροπρόθεσμα να επιδιώξουμε τους στόχους αυτούς, θα πρέπει να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που με χρονική διάρκεια περισσότερη από 18 μήνες. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η αποτροπή συγκρούσεων θα πρέπει να ενσωματωθεί με τις άλλες πολιτικές και τις άλλα μέσα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να αποδυναμωθεί με τα άλλα μέσα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ε, ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία του μέσου αυτού είναι το πόσο γρήγορο είναι για την χρηματοδότηση. Δεν είναι όμως αρκετά γρήγορο. Σε διάφορες περιπτώσεις η αρχική ιδέα του να επιτευχθεί κάτι γρήγορα μέχρι την ε, περίοδο χρηματοδότησης, μέχρι την ε, χρονική στιγμή χρηματοδότησης, διαρκεί πάρα πολύ. Άρα, οτιδήποτε επιταχύνει το μέσο αυτό θα το ωφελήσει ιδιαίτερα, θεωρώ. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δημοκρατικής εποπτείας και της ε, ταχύτητας του μέσου. Γιατί αν η δημοκρατική υποπτία καθυστερήσει ιδιαίτερα κάποια, κάποιους βραχυπρόθεσμους στόχους, νομίζω ότι αυτό θα ήταν αρνητικό. Αν και ασφαλώς μακροπρόθεσμα αυτή η υποπτία είναι σκόπιμη και θυμητή. Τώρα, ο όγκος της χρηματοδότησης έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με αυτό που είχε προτεθεί στις προηγούμενες ε, δημοσιο... δημοσιοοικονομικές αλλά είναι μικρότερο το ποσοστό αυτή τη φορά στο κεφάλαιο 4 σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Γιατί κάποια από τα υπόλοιπα μέσα αυξήθηκαν περισσότερο. Αλλά καλύτερο θα ήταν να μη μειωθεί το IFS. Επίσης υπάρχει μία πρόταση για να αυξηθεί Ε, το ποσοστό του μακροπρόθεσμου ε, σκέλους του μέσου σταθερότητας και αυτό που βλέπουμε από τις ερευνές μας ότι βασικό ε, πλεονέκτημα είναι η βραχυπρόθεσμη ταχύτητα. Ασφαλώς εφόσον υπάρχουν και μακροπρόθεσμοι στόχοι και δεσμεύσεις και γι' αυτό λοιπόν ε, συστήνουμε προσοχή σε ό,τι αφορά την αύξηση του μακροπρόθεσμου σκέλους του μέσου. Τέλος, ανακύπτει το ερώτημα της συμπληρωματιότητας και της διαφοροποίησης μεταξύ άλλων ε, μέσων όπως το μέσο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά θα πρέπει να το επανεξετάσουμε ενδεχομένω. Αλλά εν γέννη πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και ωφέλιμο ε, εργαλείο για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστεί ότι θα... Μάλλον θα πρέπει βασικά να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθούν τα θετικά του στοιχεία παρά ότι θα πετύχουμε κάτι καινούργιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μόλ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το γεγονός ότι προσκάλεσε το γραφείο για τη δημιουργία, για την οικοδόμηση ειρήνης να συμμετάσχει στη συζήτησή σας για το μέσο σταθερότητα. Δεν θέλω να κάνω μονάχα κάποια σχόλια για το τωρινό μέσο σταθερότητας και κάποια ακόμα σχόλια για το διάδοχο εργαλείο και τις επίσης τις προτάσεις που αφορούν τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να πω πρώτα ότι το δικό μας όργανο έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα το μέσο για την σταθερότητα και έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα καινοτόμε προσπάθειες για την επίτευξη τη ειρήνη. Δυστυχώ και άλλοι πιστεύουν, και κρατημέλη και διεθνεί οργανισμοί, και επομένω, είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να καταφύγουν στι υπηρεσίε αυτού του εργαλείου για τη σταθερότητα. Χαιρετίζουμε πολλέ από τι θετικέ προτάσει για το νέο μέσο σταθερότητα που περιλαμβάνουν την απλοποίηση των δομών του την αναφορά στην ε, πρόληψη των συγκρούσεων στο άρθρο 4 και την οικοδόμησή της ειρήνης, τα έκτακτα μέτρα αροχής και τη μνήα για ανάλυση κινδύνων σε σχέση με τις ε, ενδεχόμενες συγκρούσεις. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα υποστηρίξουν τα στοιχεία αυτά της νέας πρότασης. Έχουμε κάνει ορισμένε προτάσεις για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του μέσου για την ε, σταθερότητα για την πρόληψη συγκρούσεων και οικοδόμηση της ειρήνης. Αυτό αφορά δραστηριότητε βάσει του άρθρου 3 που είναι η αντιμετώπιση των κρίσεων και θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο εύκαμπτο τμήμα του μέσου για τη σταθερότητα και μπορεί να προωθήσει μια αποτελεσματική εργασία στον τομέα της οικοδόμησης ειρήνης. Υποστηρίζουμε επίση την συνιστόσα για την προετοιμασία για τις κρίσεις, του Άρθρου 4, που πρέπει να περιλαμβάνει και αυτό στοιχεία σε σχέση με την οικοδόμηση ειρήνη. Αυτό είναι το πιο καινοτόμο στοιχείο του μέσου και με ένα τρόπο με τον οποίο μπορεί να είναι πρωτοπόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να υποστηρίξει τέτοιε δραστηριότητε. Θέλουμε επίση να άρουμε την μνήμα για την αρρωγή για αποκατάσταση μεταξύ μετά από καταστροφές, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίζεται αυτό από το μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανοικοδόμηση μετά από καταστροφές. Υποστηρίζουμε επίσης τη χρήση αυτού του μέσου σε μη στρατιωτικά μέσα σταθεροποίησης. Και αυτό αφορά και την δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Δράσης. Νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναθεωρήσουμε και τη χρηματοδότηση για αυτές τις δραστηριότητες και να κρίνουμε καλύτερα την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος για την νέα πρόταση, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ειδικό ρόλος της, για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το άρθρο 5. Κατά την άποψή μας, οι παγκόσμιες και διεθνικές απειλές οι οποίες υπάρχουν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονάχα από φορεί ασφαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στι εταίρε χώρε. Τέλο, εν κατακλείδη, πιστεύουμε ότι η συνολική αποτελεσματικότητα του μέσου σταθερότητα μπορεί να αυξηθεί ιδιαίτερα με τη μεταρρύθμιση και των άλλων εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων. Και υποστηρίζουμε εδώ την υποστήριξη της ειρήνης και την ε, ε, πρόληψη συγκρούσεων όπως προτείνεται με συμμετοχή στα γεωγραφικά προγράμματα. Last Τέλος, η κυρία Ξτέσκου. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την πρωτοβουλία για την διαχείριση κρίσεων. Όπως ξέρετε, είμαστε μία ε, οργάνωση του Φιλανδική, του Πρόεδρου Πατισάρη. Το 2004 ιδρυθήκαμε και ασχολούμαστε με διάφορες περιοχές στον κόσμο. Στο Καραμπάχ, για παράδειγμα, υποστηρίζουμε την Βρετανιστερία, την υποστηρίζουμε το διάλογο στον Ιεμένη, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, τον Νότιο Σουδάν και για την εφαρμογή των project αυτό Έχουμε λάβει χρηματοδότηση από το μέσο σταθερότητα και σήμερα μου ζητήθηκε να μιλήσω σε ό,τι αφορά τι εμπειρίε μα από την εφαρμογή του μέσου και θα σα μιλήσω ιδιαίτερω για το τι διαπιστώσαμε με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία σε ό,τι αφορά το project του Ναγκόρνο Καραμπάγα που χρηματοδοτείται από το μέσο σταθερότητα. Διάφορα στοιχεία ήθελα να αναφέρω, ωστόσο θα περιοριστώ σε τέσσερα. Καλώς ορίζουμε καταρχάς την πρόταση να επιταχυνθεί η χρήση και η εφαρμογή του μέσου και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπογραμμιστεί περαιτέρω η απλοποίηση των κανόνων για την παροχή τέτοιας βοήθειας το EPNK έχει ε, ωφεληθεί από την υποστήριξη 18 μηνών 2010 μέχρι 2011 και όπως θα ξέρετε είναι μακρά η σύγκρουση στον Αγκόρνο Καραμπάχ και 18 μήνες δεν ε, αρκούν για την υποστήριξη της ειρήνης στην περιοχή. Έχουμε υποβάλει αίτημα τον Ιούλιο του 2011 για να συνεχίσει η χρηματοδότηση, για να συνεχίσουμε τις δραστηριότητε μας, αλλά δεν έχουμε ακόμα λάβει απάντηση. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτή χρειάζεται για την συνέχιση των δραστηριοτήτων μας και πρέπει να πω ότι αυτή η αβεβαιότητα έχει ε, αρνητικό αντίκτυπο στο project και δυστυχώς πρέπει να πω ότι η εικόνα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τυπικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του EPNK ε, είναι αρνητική. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο ήθελα να τονίσω σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 και πάλι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα έκτακτα μέτρα και τα προσωρινά μέτρα να μπορούν να έχουν διάρκεια έως και 13 μήνες σε τέτοιες ε, συγκρούσεις παρατεταμένες όπως τον Αγκόρνο Καραμπάχ ε, όπου χρειάζεται υποστήριξη Προ την ε, κοινωνία των πολιτών. Γιατί συστημικέ αλλαγέ από βραχυπρόθεσμα προγράμματα δεν πρόκειται να προκύψουν. Και όπω ξέρετε, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση από το EEPI ή από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε το άρθρο 7 και την αλλαγή που επιφέρει. Τρίτο σημείο που ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με το θέμα του συντονισμού, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το άρθρο 2 που αναφέρεται στη συμπληρωματικότητα και στη συνεκτικότητα της αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε ότι είναι ουσιώδες. Ιδιαίτερα όταν εφαρμόζει ε, τέτοια έργα σε πολύ ευαίσθητα περιβάλλοντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε περιφερειακές συγκρούσεις που ενδεχομένως να διαδοθούν και σε άλλες χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού σε διάφορες περιπτώσεις μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Και βρισκόμαστε ως μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε μια θέση που αναγκαζόμαστε να συντονίσουμε ε, το έργο αυτό. Για παράδειγμα, στο EPNK, στα πλαίσια της Γεωργία, επηρεάζει και την Αρμενία, το Ζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες. Επίσης ήταν πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναμειγνύεται και να συμμετέχει πιο πολύ στη φάση του προγραμματισμού Όπως είπε και ο συνάδελφος, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχει πιο πολύ στον προγραμματισμό και να συνεργάζεται πιο πολύ με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σημείο για την αξιολόγηση. Εμείς, για παράδειγμα, έπρεπε να αξιολογήσουμε μόνοι μας το πρόγραμμα και δεν θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής αξιολόγησης γιατί αυτό δεν μπορεί να τροφοδοτήσει ε, το πρόγραμμα. Δεν μπορούν τα αποτελέσματα αυτά να εισέλθουν και πάλι στο πρόγραμμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνεται από την υπηρεσία εξωτερική δράση αυτή <coughs> η αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Η συγκήτρια, κυρία Μπράντνερ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω και τους τέσσερις εμπειρογνώμονους μας και σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια και τη στιγμή που έχετε αναφερθεί στα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Θέλω απλώς να σταθώ σε ορισμένε από τις παρατηρήσεις σας και να κάνω κάποια σχόλια στην αρχή σε σχέση με τον τίτλο του μέσου αυτού. Λέγεται μέσο για σταθερότητα. Αλλά η σταθερότητα έχει πάρει μια κάπως αρνητική χρειά στη Βόρεια Αφρική, γιατί για τις χώρες αυτές δίνει την εντύπωση ότι θέλουμε απλώς να κρατήσουμε τους δικτάτορες στη θέση τους. Πολλέ χώρε λοιπόν όπου χρησιμοποιούμε το μέσο σταθερότητος έχουν γίνει σκεπτικοί στρίες για τα θέματα αυτά και καταλαβαίνω ότι αυτή η απόχρωση τη σταθερότητα είναι λίγο αρνητική για την περιοχή αυτή. Θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα λοιπόν το μέσο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κρίσεων, γιατί για αυτό το θέμα αναφέρεται αυτό το εργαλείο. Μπορούμε να εξετάσουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα αλλαγή του τίτλου. Δεύτερον, εμβέλεια αυτού του μέσου. Νομίζω ότι αναφέρθηκε δύο φορές ότι υπάρχει μια επικάλυψη μεταξύ του μέσου σταθερότητα, όπως προβλέπετε τώρα, και το φορέ για ανθρωπιστική βοήθεια. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε και περισσότερη σαφήνεια και λιγότερη επικάλυψη, ιδίω όταν δεν έχουμε επαρκή πόρου, Αλλά όταν έχουμε ε, κινδύνους ασφαλείας μετά από φυσικές καταστροφές, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Μέσα από την ανθρωπιστική βοήθεια. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να διατηρήσω το μέσο για τη σταθερότητα μονάχα σε τομείς που έχουν να κάνουν με προβλήματα ασφάλειας και όχι σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Τρίτο σημείο που αναφέρθηκε και αυτό, το θέμα της συμμόρφωσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια των μέτρων κατά της τρομοκρατίας. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω αυτό το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν όπως ξέρετε, ο Επίτροπος Φερχόβεν κάποια στιγμή είχε υπογράψει μία δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών μέτρων, αλλά ποτέ δεν αναπτύχθηκαν κατευθυντήρες γραμμές οι θεσμικοί μηχανισμοί για να εφαρμοστεί αυτή η ρήτρα από την κυρία Φερεροβάλτερ που ήταν τότε αρμόδια επίτροπος ή την κυρία Άστον που είναι τώρα αρμόδια. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, Αντίστοιχε κατευθυντήρες γραμμές από το αγγλικό Foreign Office και ίσως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα και να ζητήσει σε μια δήλωση να εφαρμοστούν μηχανισμοί παρακολούθησης ανθρωπίνων των δικαιωμάτων εμπνεόμενοι από τις κατευθυντήρες γραμμές του Foreign Office, του Υπουργείου Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης θα ήθελα να υπάρξει και μια μεγαλύτερη μνήμα στην έννοια του διαλόγου για τη διαμεσολάβηση σε κρίσεις και επίσης πάλι θέλω να τονίσω το ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να εξάρω ιδιαίτερα το ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εξπόστη αξιολόγηση. Γιατί συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να έχει κανείς μια άποψη εκ των, προτέρων γιατί μιλάμε για ταχείες διαδικασίες αλλά τουλάχιστον στο επίπεδο της εκ των υστέρων αξιολόγησης θα μπορούσε να έχουν ένα κομβικό ρόλο οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικός αυτός ο ρόλος και είναι κάτι το οποίο πάντα το διεκδικούμε σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της οκίτητος της δράσης μας, αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με τα θέματα της δημοκρατικής ε, υπολογότητος και λογοδοσίας, αλλά περισσότερο με τον οικονομικό έλεγχο. Από τον τριγωνικό διάλογο για τον δημοσιονομικό κανονισμό είναι δυστυχώς κρίμα που η ευκαμψία που ζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καλύτερη πρόληψη των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των κρίσεων δεν έγινε δεκτό από το Συμβούλιο. Δεν είναι βέβαια δικό μα ρόλο να αποφασίσουμε. Εμεί είχαμε μια καλή θέση ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διευκολύνουμε αυτού του μηχανισμού που θέλατε και να είναι πιο γρήγορη η λειτουργία του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά αυτό μα το εμπόδισε το Συμβούλιο. Δεν πιστεύω όμω ότι το τμήμα του δημοκρατικού ελέγχου θα πρέπει να επιβραδυνθεί περισσότερο. Τέλος, για, το, για τη συνολική χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι το μέσο ε, σταθερότητας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την ταχύτητα αντίδρασής του. Γι' αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε στα προηγούμενα ποσά χρηματοδότησης, αλλά φυσικά όλα εξαρτώνται και από την ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αυτού του μέσου. Αν διευρυνθεί και σε θέματα φυσικών καταστροφών και δημόσια υγεία πρέπει να έχει και μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Πάντως ευχαριστώ πολύ του ε, εμπειρογνώμου και περιμένω τώρα τα ερωτήματα των συναδέλφων μα και την άποψη τη Κομισιόν Allora, prima intervenire sarà il relatore Πρώτα ο συνάδελφο Γουαλτιέρη που είναι ο σκιώδης εισήγητή, και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι ο Σκιώδης εισηγητής για τη σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ τους εισηγητές που μας ε, έδωσαν ένα πλαίσιο εξωτερικό πλαίσιο αξιολογήσεων για αυτό το μέσο, το οποίο είναι ένα μέσο πάρα πολύ σημαντικό. Και για διαδικαστικούς λόγους και για ουσιαστικούς λόγους. Σημερίζομαι τις θέσεις ουσίας της εισηγήτριας. Η θέση, η έκθεση συνολικά είναι δεκτή. Υπάρχουν μερικά εκκρεμή ζητήματα που πρέπει, στα οποία πρέπει να εμβιαθύνουμε. με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η πρόταση εισάγει αλλαγές, άλλες καλές, άλλες όμως ε, συζητούμε, αμφιλεγόμενες, αλλά κατά βάθος όμως είναι και πολύ συντηρητική. Διότι η βάση αυτής της πρότασης θυμίζει μία πρόταση προ-Λισαβόνας θυμίζει το παλιό μέτρο. Τα άρθρα 3, 4 και 5 άλλαξαν ε, ως προς τον τίτλο για το peace building, αλλά στο άρθρο 1 λέμε ότι στόχος είναι να διευρύνουμε τα μέσα ανάπτυξης και συνεργασίας της Ένωσης. Μας παραπέμπει δηλαδή σε μια άλλη τοποθέτηση. σε τομεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παλιά ήταν κατακαιρματισμένοι αλλά σήμερα είναι ενωμένοι και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Για άλλα ζητήματα, όπως είπε και η συνάδελφος Μπραντνερ, έχουμε κάποιες κριτικές, πιο συγκεκριμένα για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όχι μόνο για το θέμα των εντεταλμένων πράξεων, ε, για τη μείωση πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει του άρθρου 7, 7.7 είναι πιο περιορισμένη ενημέρωση από ό,τι στον προηγούμενο κανονισμό. Επίσης, στη βάση όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπόψη η νέα συνθήκη αλλά δεν λαμβάνονται και άλλα νέα πλαίσια τα οποία έχουν διαμορφωθεί όπως το CFSP. Δεν υπάρχει σαφήνεια. Σύμφωνο με αυτά που είπαν μερικοί από τους εισηγητές ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την ιδιαιτερότητα αυτού του μέσου σταθερότητας και να ενισχύσουμε τις ε, να σταθεροποιήσουμε αυτές τις ενιαίες θέσεις χωρίς να έχουμε υπαστή μέτρα. Για τους 30 μήνες πρέπει να το σκεφτώ. όπως ε, και την ε, διατύπωση για την εισαγωγή στο παράρτημα του άρθρου 4 των ε, κλιματικών ιδιαιτεροτήτων που πρέπει να επισέλθουν στην ιδιαιτερότητα αυτού του μέσου. Επιφυλάσσομαι λοιπόν να το σκεφτώ και να λάβω υπόψη μου και τη συζήτηση σήμερα για να καταθέσω τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να θέσω κάποια ερωτήματα και θα τα παρουσιάσω αυτά από πλευρά μου, αλλά και εξ ονόματο του κυρίου Κέλαμα ο οποίο μου ζήτησε να μιλήσω εξ ονόματο του. Καταρχά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά του συμπεριγνώμονε. Και αυτά που είπαν για το ΙΕΦΕΣ. Ορίζεται εξίσου ξεκάθαρα όσο σήμερα σε ό,τι αφορά το σύνδεσμο με τα άλλα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς προκειμένου να υπάρχει επαρκή συντονισμός και σύνδεση μεταξύ των οικονομικών μέσων. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες το εξής. Ποια είναι η άποψή τους σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί νομίζω ότι διαπιστώνουμε ότι το IFS ε, αποτυπώνει την ε, λογική της ε, συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε και θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης. Άρα η συνεκτικότητα εξαρτάται από τις ε, δράσεις στις οποίες πρόκειται να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη και το πόσο αντιδρούν σε καταστάσεις κρίσης ε, ή αποτροπή συγκρούσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους εμπειρογνώμονες τι πιστεύουν ότι θα πρέπει να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξ ονόματο του κυρίου Κέλλαμ θα ήθελα να πω τα εξή. Δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εδώ πέρα για να θέσει τα ερωτήματά του. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους εμπρεγνώμονες για το άρθρο 8 τμήμα 2 σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών που αναφέρεται στο σημείο αυτό και τη δυνατότητα να, οριστεί, να οριστούν κάποια benchmarks για τη συμμετοχή αυτή. ορίζονται με σαφή τρόπο σήμερα ή πιστεύουν οι εμπειρογνώμονε ότι θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη αναφορά στην κοινωνία των πολιτών. Μία άλλη ερώτηση τώρα από τον κύριο Κέλαμ. Για το παράρτημα 1, τμήμα D, δέλτα, για την υποστήριξη των διεθνών δικαστηρίων, των διεθνών ποινικών δικαστηρίων. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για το άρθρο αυτό. Ο κύριος Λάμστορφ, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο οδηγίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω μονάχα με ορισμένες απλές παρατηρήσεις. Εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο νομικό εργαλείο, ένα μάλλον ε, ειδικό πολιτικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα πρέπει να ασχοληθεί με θέματα τα οποία δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η συγκατάθεση μιας χώρας στην οποία θα λειτουργήσει αυτό το μέσο και αυτό ε, επιτρέπει βέβαια και με μεγαλύτερη ευκαμψία σε αυτό το μέσο, αλλά μπορεί να αποτελέσει και μία, ένα ασθενές στοιχείο, διότι λόγω αυτής της ταχύτητος δράσης εναντί των άλλων ε, ε, εργαλείων δεν θα μπορεί να τον καλύψει ενδελεχώ, αλλά το γεγονό ότι μπορεί να έχει ταχεία δράση, αυτό καλύπτει κενά από τα άλλα μέσα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όμω είναι να εξασφαλίσουμε καλύτερα ποια είναι τα όρια του πεδίου εφαρμογή του μέτρου αυτού. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το οποίο προτείνει η συγγήτρια, να παραμείνουμε μονάχα στον τομέα της πρόληψης των κρίσεων και της οικοδόμησης ειρήνης και μόνο. Κατά την άποψή μου αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα από το να διευρύνουμε αυτήν την εντολή. Εκεί που δεν είμαι τελείως σίγουρος είναι πώς θα εξασφαλίσουμε να έχουμε μια στρατηγική αντιμετώπιση, μια πλήρη αντιμετώπιση, ενώ συγχρόνως αυξάνουμε την ικανότητα αντίδρασης αυτού του εργαλείου. Θέλουμε από την αρχή να έχουμε μια γρήγορη αντίδραση και να αντιμετωπίσουμε την αντίφαση μεταξύ της ταχείας αντίδρασης και της στρατηγικής αντιμετώπισης σε σχέση με τον τίτλο. Εγώ είμαι έτοιμος να υποστηρίξω οποιαδήποτε ε, ονομασία. Δεν έχω κάποιο φετίχ με τη λέξη σταθερότητος και γνωρίζω ότι πράγματι έχουν προκύψει κάποια προβλήματα λόγω της αραβικής ε, άνοιξης. Εγώ δεν έχω τώρα την ίδια αντιμετώπιση όπως είχε ο Τζος Μπούς, ο οποίος Μιλούσε για τη δημοκρατία και επομένω πήρε άσχημο όνομα η δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε αλλαγή. <clears throat> Βρίσκω θετικό ότι και η ομάδα μου το ίδιο, ότι η απλοποίηση των διαδικασιών λαμβάνεται και αυτή η υπόψη και επίσης και η ευκολότερη πρόσβαση για τους δικαιούχους, τους δυνητικούς Όλα αυτά λοιπόν γενικά θα ευνοήσουν τους στόχους αυτού του νομοθετήματος για τα έκτακτα μέσα υποστήριξης. Υπάρχουν τώρα τρία σημεία στα οποία εγώ θα καταθέσω κατά πέσα πιθανότητα τροπολογίες μαζί με την πολιτική μου ομάδα. Πρώτα σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την πρόληψη κρίσεων και για τις ε, παγκόσμιες και δια, ε, δια, απειλές εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα με ποιο τρόπο καθορίζουμε την έννοια του συντονισμού και πώς θα συντονίζεται αυτό το εργαλείο με συμπληρωματικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει ο συντονισμός να μείνει σε ένα θετικό επίπεδο. Ένα τρίτο σημείο φυσικά υπάρχει είναι και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν διαφωνώ καθόλου με την εισηγήτρια γιατί και για τη δική μας ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και πρέπει να, να αναλάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Η ε, κυρία Μουνής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ στους εμπειρογνώμονες που μας ενημέρωσαν για τις αλλαγές ε, στο μέσο σταθερότητα. Έχω ορισμένε ερωτήσεις. Εγώ συντάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών για αυτό το θέμα και συμμερίζομαι με την κυρία, αυτά που είπε και η κυρία Μπραντνερ και η κυρία Λάμστορφ Λοιπόν, πρέπει να ε, διασαφιστεί σαφώς το θέμα των ενταλμένων πράξεων για το Κοινοβούλιο και για τις νέες προτεραιότητες για το μέσο σταθερότητας και πιο συγκεκριμένα για την ασφάλεια και για την διακίνηση φαρμάκων μαϊμού. Δεν ξέρω πώς εμείς μπορούμε να δώσουμε ε, να το ε, περιεχόμενο σε αυτό το μέσο όταν ε, δηλαδή το στρεβλώνουμε με μέτρα τα οποία δεν έχουν να κάνουν ούτε με τη σταθερότητα ούτε με το peace building. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν και να μου το πει η Κομισιόν η κυβερνοασφάλεια αν θα πρέπει να είναι ε, μέσα στο αντικείμενο αυτού του μέσου όπως επίσης και η διακίνηση φαρ, ε, φαρμάκων μαϊμού. Σίγουρα η διακίνηση φαρμάκων μαϊμού ε, είναι επιβλαβής ε, για το, τους πληθυσμούς διαφόρων ε, χωρών, αλλά υπάρχουν χιλιάδες απειλές κατά της υγείας ή κατά των πληθυσμών με σε διαφορετικές συγκυρίες η δημοκρατική σταθερότητα, η βοήθεια των πληθυσμών κατά τις φάσεις ε, κρίσης ε, είναι η ουσία αυτού του μέσου, όχι όλες οι άλλες απειλές ε, που έχουμε σε, μια, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δεν πρέπει εμείς να το υπερφορτώσουμε αυτό το μέσο. Και επίσης αναρωτιέμαι αν δημοσιονομικά στέκει να φορτώσουμε με νέες αρμοδιότητες αυτό το σχέδιο. Εγώ θα ήθελα να ξέρω για αυτές τις νέες προτεραιότητες που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο του, μέσου σταθερότητας. Τι χρηματοδότηση έχουν, τι προβλέπετε στον προϋπολογισμό γι' αυτό. Εγώ θέλω διαμεσολάβηση peace ε, building, ε, δημοκρατικά θεσμικά όργανα και ενίσχυσή τους, αυτά που είχαμε δηλαδή στο παρελθόν ως προτεραιότητες, όχι όλα αυτά τα καινούργια. Ευχαριστώ. Ωραία. Η κυρία Τζέννη. από την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Ένας βασικού στόχους είναι η οικοδόμηση τη Ειρηνή. και αυτό προέρχεται από το γεγονό ότι τα πιο πολλά παραδοσιακά μέσα ε, σκοπό έχουν να υπάρχει αποτελεσματικότητα στο κόστο. και έτσι το κίνητρο είναι να δαπανώνται πολλά χρήματα για να περιοριστεί το ε, γραφειοκρατικό άκτος. Ξέρουμε όμως ότι σε περιπτώσεις σύγκρουσης είναι τα πολύ, ένα πολύ μικρό ποσό χρημάτων μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διακριτικοί παράγοντες που θα ε, λειτουργήσουν από την κοινωνία των πολιτών. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό πλεονέκτημα του μέσου σταθερότητα. Ε, δυνατότητα χρηματοδότησης μικρών project, μικρών έργων μέσω της κοινωνίας του πολιτών και με δυνατότητα ευελιξίας. Αυτός ο νέος κανονισμός νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και γι' αυτό τον υποστηρίζουμε ιδιαίτερος. Θεωρούμε ότι οι προτάσεις κινούνται στην κατεύθυνση του να εφαρμοστούν οι φιλοδοξίες της συνθήκης της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά και το άρθρο 21. Σα Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βιλανόβα. Νομίζω ότι το πλεονέκτημα του μέσου σταθερότητα είναι ότι αντιμετωπίζει θέματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κανένα άλλο μέσο. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ε, δίδεται και εγγυάται και την επικουρότητα. Και αυτό πλέον ε, κατοχυρώνεται και στον κανονισμό. Δεν αναφέρονταν προηγουμένω. Για πρώτη φορά, λοιπόν, αναφέρεται ότι η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από άλλα μέσα. Αυτό είναι κριτήριο ε, για την παροχή της χρηματοδότησης. Ε, τέσσερις όροι υπάρχουν. Καταρχάς, ε, όταν θα χρειάζεται ταχεία απάντηση σε μία κρίση. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, υπάρχει μία απειλή υπερεθνική. υπερεθνική που εξορισμού ξεπερνάει τα όρια ενός εθνικού εργαλείου όπως το DCI, το MPI και το καθεξής. Ε, ένα παράδειγμα. Ε, με κοκαίνη και τράφικιν κοκαίνης, ε, παράνομη διακίνηση ε, κοκαίνης από την Λατινική Αμερική μέσω της Αφρικής ε, στην Νότιο Ευρώπη. Όπως βλέπετε, κανένα γεωγραφικό εργαλείο δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο αυτή την απαλή. Και αυτό το βλέπουμε λοιπόν ε, ότι παρουσιάζεται συχνά. Αυτό λοιπόν είναι το πλεονέκτημα. Μία άλλη περίπτωση όπου για παράδειγμα ε, πρέπει να υποστηρίξουμε δράσεις κατά της τρομοκρατίας. Να σας υπενθυμίσουμε και το DDF και το DCI που είναι αναπτυξιακά μέσα έχουν συγκεκριμένους όρους τους οποίους ε, είναι δεσμευτικοί. Το όργανο για τη δημοκρατία. Το εργαλείο για τη δημοκρατία. Και υποστηρίζουμε την ανάπτυξη πολιτικών ε, για την οικοδόμηση ειρήνης ε, που δεν έχει να κάνει ιδιαίτερα με κάποια χώρα σε ό,τι αφορά στα πλαίσια της ΕΠΛΟ, για παράδειγμα που δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν χρηματοδότηση από, άλλες, ε, από άλλα μέσα. Είναι σαφής λοιπόν η προστιθέμενη αξία και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε ακριβώς να τονίσουμε τις τέσσερις αυτές τις περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας θα θέλαμε να τονίσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το οποίο ε, ανέφεραν και οι δύο εμπειρογνώμονε και η κυρία Μπρνάντνερ. Από ό,τι ξέρετε, τονίζουμε ιδιαίτερα την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω υποστήριξης, για παράδειγμα, στην προσχώρηση στην εφαρμογή μέσων των ΟΗΕ ή άλλων διεθνών οργανισμών, προωθώντας επίσης ε, μια αστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε σχέση με αρχιωτικές μεθόδους και ε, υποστηρίζοντας ε, τον δημοκρατικό έλεγχο. Και ένα από τα καινούργια στοιχεία του κανονισμού είναι ότι αναφέρουμε συγκεκριμένα το ρόλο των κοινοβουλίων ως αρμόδια όργανα για την εποπτεία του μηχανισμού ασφάλειας του κάθε κράτους. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητες ε, τις αντιτρομοκρατικές. Ε, για παράδειγμα, πέρσι η κυβέρνηση της ε, αντέδρασε βία σε μία σύγκρουση, σε μία ε, σε ένα ξεσηκωμό, αποφασίσαμε να σταματήσουμε την χρηματοδότηση. Ο κύριος Ντόιλ είναι ο πρώτος ομιλητής της Κομισιόν. Oh, uh, Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιχαήλ Δόιλ από την Υπηρεσία του Μέσου Εξωτερικής Πολιτικής κάποια σύντομα σχόλια για ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία ηγέτησαν το θέμα της ταχύτητας καταρχήν. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα, πολύ πρόσφατο πριν από δέκα μέρες, τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει έκτακτη βοήθεια για να ξεκινήσουμε την αποστολή παρακολούθησης στη Συρία. Μέσα σε μία εβδομάδα έγιναν συζητήσεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ολοκληρώθηκε μια δέσμη αποφάσεων και μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες, είχαμε καταφέρει μέχρι σήμερα το πρωί να πάρουμε αποφάσεις και σήμερα το απόγευμα έγινε η, θα γίνει συμφωνία για την ε, αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και ελπίζω ότι όλα αυτά θα είναι έτοιμα την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά θα, δείξουν, θα επιτύχουν το να λειτουργήσει αυτή η αποστολή με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό δεν το κάνουμε κάθε μέρα είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά όταν μας πιέσουν μπορούμε πράγματι να το κάνουμε. Πολλές φορές χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να καθορίσουμε τι μορφή θα πάρει η παρέμβασή μα. Για το θέμα τη συμπεριληψη, της δυνατότητα υποστήριξης για φυσικές καταστροφές. Ε, άκουσα αυτά τα οποία είπε η συγγήτρια σήμερα το απόγευμα για τα θέματα αυτά, αλλά και πάλι θέλω να σα δώσω κάποια παραδείγματα όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την πρόσθετη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε τέτοιε καταστάσει. Η ΑΙΤ μετά από το σεισμό ή το Πακιστάν μετά τι μεγάλε πλημμύρε πριν από 2-3 χρόνια. Ήταν απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα στι χώρε αυτέ και για να γίνει αυτό έπρεπε να δει ο πληθυσμό ότι έχετε κάποια ανακουφιστική βοήθεια. Όχι μόνο η άμεση ανακουφιστική βοήθεια, αλλά και αυτή η οποία βοηθάει τι πρώιμε προσπάθειε ανοικοδόμηση. Και ήταν το μόνο εργαλείο το οποίο μπορούσε να λειτουργήσει. Όπω είπε και ο κ. Λάμστορφ, είμαστε πάντα ένα εργαλείο τελευταία καταφυγή. Αλλά μπορούμε πάντα να συνεργαστούμε με του συναδέλφου μα αν υπάρχουν και άλλα μέσα. Εμεί προσπαθούμε πάντα να κάνουμε γρήγορα τα πράγματα και αυτό έχει σταθεροποιητικό αποτελέσμα η Δομινικανική Δημοκρατία που είχε πολλούς ε, πρόσφυγες από την Αιτή δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της το ΕΤΑ για τους πρόσφυγες αυτούς. Αλλά αν δεν υπήρχε βοήθεια θα υπήρχε μεγαλύτερη αναταραχή στη χώρα αυτή. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση στο ΕΤΑ και επομένως το, ε, η επόμενη μέρα <clears throat> της φυσικής καταστροφής αντιμετωπίστηκε. Χαίρομαι για το γεγονός ότι υποστηρίζετε τις ε, προτάσεις για ευελιξία που έχουμε προτείνει στο νέο κανονισμό. Τα περισσότερα στοιχεία ήρθαν από, τον οριζόντιο, από την οριζόντια αξιολόγηση που έγινε πρόσφατα, που περιλαμβάνει τα μέτρα άμεσης ε, υποστήριξης, που περιλαμβάνουν και περιοχές όπως τον Αγκόνο Καραμπάχ. Η ιδέα του να περάσουμε στους 30 μήνες χωρίς εξαιρέσεις είναι λοιπόν πολύ θετική. Κατανοούμε αυτά που λέτε για την αξιολόγηση των σχεδίων είναι στο μέσο που κάνουμε περισσότερα πράγματα για να αναπτύξουμε μια καλύτερη προσέγγιση. Για τα διεθνή δικαστήρια έχουμε δώσει ουσιαστική <clears throat> υποστήριξη. Είμαστε το μόνο μέσο που μπορεί να κινητοποιηθεί για τα διεθνή δικαστήρια και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητας. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ πέρα. Mr. Meyer. Ο κύριος Thank you, Mr. Ευχαριστώ ναι, και συγγνώμη για την πρώτη φορά που ήρθα εδώ πέρα. Δεν έχω τόσα πολλά να προσθέσω σε αυτά που είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Οι να σας ευχαριστήσω για τις καλές παρατηρήσεις που λάβαμε και για την καλή, ε, τις καλές, τα καλά σχόλια. Επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις για τις νέε δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμάκων. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Αφρική, μια νέα απειλή που αφορά ιδιαίτερα την Αφρική και μπορεί να έχει πολύ αποσταθεραπευτικό χαρακτήρα και ασφαλώς και ε, τροφοδοτεί άλλου είδους εγκληματικές οργανώσεις και κυκλώματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρξει καλύτερη θεώρηση και προβολή των δραστηριοτήτων αυτών που συχνά ε, διενεργούνται από τις ίδιες ομάδες. Όπως είπατε, Υπάρχουν και οι φυσικές ε, καταστροφές που περιλαμβάνονται πλέον. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιφέρειες, ίσως και ήπειροι ολόκληροι, όπου γίνεται επένδυση μόνο στην άμυνα της ε, χώρας. Αυτό ε, είναι πολύ ακριβό και για την ίδια τη χώρα τέτοιες περιπτώσεις. Αν υπάρχει μια βιολογική φυσική καταστροφή λόγω τρομοκρατικής επίθεσης, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα στον κόσμο είναι τα ίδια. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, υπάρχουν μολύνσεις, ε, λοιμώξεις που επηρεάζουν όλο τον πληθυσμό. Αν καλυφθούν και οι φυσικές καταστροφές, και απειλές, επιθέσεις τρομοκρατικής φύσεως, νομίζω ότι είναι πιο ε, σημαντικό, γιατί ουσιαστικά ο ίδιος ο αντίκτυπος ε, προκύπτει και από τις δύο επιθέσεις και τα δύο μέσα. Επίσης ε, και στις δύο περιπτώσεις τα ίδια μέσα χρησιμοποιούνται. Άρα ίσως να είναι περιοριστικό το ότι να διευκρινίσουμε ότι πρέπει να πρόκειται υποχρεωτικά για τρομοκρατικέ επιθέσεις. Ρωτώ τώρα. Ποιος από τους εμπειρογνώμονες θέλει να απαντήσει. Ένα λεπτό. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. I would... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι είναι μοναδικό αυτό το εργαλείο για μας και θα σας έδωσα πάλι το παράδειγμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να συλλειτουργήσουμε σε αυτή τη σύγκρουση χωρίς αυτό το εργαλείο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υποστήριξη από μέσα όπως το MPI και είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από κράτη-μέλη γιατί αυτή είναι μια σύγκρουση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπλέκεται και υπάρχουν κράτη-μέλη της τα οποία εργάζονται μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ειρήνευσης. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν αυτό και το μέσο για τη σταθερότητα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτό. Η άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω αφορά το θέμα που έθεσε ο κύριος Πρέντα σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Κατά την άποψή μου, το άρθρο 8 θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, γιατί λέει θα πρέπει όπου είναι απαραίτητο να γίνονται διαβουλεύσεις. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν λειτουργούμε εν κενό αέρα, λειτουργούμε σε πάρα πολύ ευαίσθητες συνθήκες μέσα σε συγκρούσεις και επομένως η διαβούλευση με τους τοπικούς εμπλεκομένους σε πολιτικό επίπεδο και την κοινωνία των πολιτών πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ προσεκτικά σαν τμήμα μια στρατηγική. Δεν μπορεί να γίνει αυτόνομα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε σχόλιο. Το άλλο το οποίο θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με το θέμα του συντονισμού. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ο συντονισμός με τα κράτη-μέλη σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα τέτοιο, κάτι τέτοιο. Στη, Μολ, στη Μολδαβία, παραδείγματος χάρη, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντονίζει την αρρωγή σε τοπικό επίπεδο. <clears throat> το πρόβλημα όμως με τον αγώνο Καραμπάχ ότι δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν τρεις εμπλεκόμενες αντιπροσωπείες Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν. Και είναι πολύ δύσκολος ο συντονισμός. Είχαμε ένα σύστημα με διοικούσες επιτροπές όπου γινόταν μια τέτοια μορφή συντονισμού. Έχει λειτουργήσει πολύ καλά το σύστημα αυτό και θα είναι καλό δεκτό για να επαναληφθεί με κάποιο εστιακό σημείο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σερίφ. πάρα πολύ σύντομα, καταρχήν είχε σχέση με την, το συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Αν έχετε καλή ανάλυση σε σχέση με τη σύγκρουση, τι γίνεται σε μια περίπτωση το οποίο την χάνει κοινή αντιμετώπιση και κοινή στρατηγική αντιμετώπιση τη κρίση από τα κράτη-μέλη, τότε είναι πολύ καλύτερη βάση συντονισμού από το να αντιμετωπίζει κανεί μονάχα σαν εργαλείο το φορέα αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα, ένα ευρύτερο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο ερώτημα τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνθήκε κρίση ή συγκρούσεων για να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, μεταξύ των οποίων και το μέσο για τη σταθερότητα. Πώ μπορούν να συμμετάσχουν λοιπόν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση αυτού του θέματο και φυσικά πρέπει να σκεφτούμε και για τον ρόλο των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση επιτοπίω. <clears throat> για το θέμα του αν είναι οι δημοσιονομικοί κανονισμοί ή η κατεξουσιοδότηση πράξη δυνητικά που θα τροχοπεδίσουν τη διαδικασία, εγώ συμφωνώ με την κυρία Μπραντνερ ότι κυρίως είναι οι δημοσιονομικοί κανονισμοί οι οποίοι οδηγούν σε μια βραδιπορία. Και, και οι υπάλληλοι που τα διαχειρίζονται τα κονδυλευτά και οι αποδέκτες θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Τα παραδείγματα που διαλέξαμε όταν κάναμε την αξιολόγηση μας έκαναν απόλυτα σαφές ότι ήταν πολύ δύσκολο για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν τα θέματα αυτά, αλλά τους ποδηγετούσε, τους έδαινε χεροπόδαρα ο κανονισμός τον οποίο πρέπει να τηρήσουν. Κύριε Μαρτινέλη, ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνδέσω το τελευταίο σημείο αυτό του Άντριου και το πόσο εύκολο είναι να διαδημηθούν οι πόροι. Να σας πω ότι από την εμπειρία μου στην Αφρική για τα CSDP πρέπει να σας πω ότι δεν είναι εύκολο να δοθούν χρήματα, να δοθούν πόροι σε ό,τι αφορά τέτοια project. Επικοινώνησα τότε με το υπεύθυνο για το IFS και μου αναφέρθηκε ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούσαν ακόμα να διανεμηθούν γιατί είχαν ήδη προγραμματιστεί σε ό,τι αφορά τώρα τις, ε, τα μικρά ποσά που διανέμονται. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν γίνεται πάντα με συνεκτικό τρόπο και νομίζω ότι η έμφαση είναι μάλλον πιο πολύ στο να μειωθούν τα γραφειοκρατικά βάρη παρά ε, το να ανταποκριθούμε σε πραγματικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τον προορισμό των, των χρημάτων. Το θέμα των μέτρων ε, συμφιλίωσης ε, είναι σημαντικό, αλλά αμφιβάλλω κατά πόσον η αντιπροσωπεία έχει την ικανότητα να ορίσει τους τομείς όπου μπορούν να διανεμηθούν τέτοια κονδύλια μέσω διαμεσολάβησης, γιατί λίγοι από τους υπεύθυνους ε, του EFSF έχουν τέτοιες ικανότητες. Σε ό,τι αφορά τα benchmarks, να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζω, η, πολιτεία, η κοινωνία των πολιτών δεν ε, συμμετέχει σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και τον ορισμό των benchmarks. Και συμφωνώ ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί και το σκέλος της αξιολόγησης. Και τώρα ο λόγος στην εισηγήτρια για να εξαγάγει συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις ερωτήσεις που έθεσαν στους εμπειρογνώμονες και ευχαριστώ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν να ε, συγχαρώ τον κύριο Ντόλ για την ταχύτητα του πακέτου για τη Συρία. Κύριε Λάμσδορφ, λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ισορροπία αφενός μεταξύ ευελιξίας και αφετέρου να μην καταστεί και πάρα πολύ εύκολο στη χρήση αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο. Και είναι φυσικά δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία. Ευχαριστώ τον Μαριόν για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της για τη χρηματοδότηση των έργων και ποιο είναι το πλεονέκτημα για τον κύριο Γκουαλτιέρη που αναφέρθηκε στην αλλαγή του κλίματος. Δεν νομίζω ότι πολλοί πράσινοι εισηγητέ θα συμφωνούσαν όπως εγώ να αφαιρεθεί αυτή η αναφορά. Μπορούμε να το σκεφτούμε περαιτέρω όμως το θέμα αυτό. Να επανέλθω στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σαν συντομία, κύριε Ντόιλ, Αναφερθήκατε στην Δομινικανή Δημοκρατία και για το EDF που δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τους πόρους για τους πρόσφυγες. Ε, δεν ε, είναι επαρκής αυτός ο λόγος. Λυπάμαι. Δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι α, δεν θέλουμε να, απλά να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους αυτούς. Θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει κάποια άλλη πηγή για τους πόρους αυτούς. Δεν μπορώ να αυτό που έχω υπόψη μου είναι ότι τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς και όχι τόσο πολύ για ανθρωπιστική βοήθεια, για ανοικοδόμηση. Συμφωνώ με αυτό που είπατε για τα μικρά ποσά. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς συνδέεται και με το προσωπικό, τον αριθμό του προσωπικού που έχουμε στη διάθεσή μας στο Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί όταν ζητάμε πιο πολύ πιο πολλά μικρά ποσά θα πρέπει να ζητάμε και πιο πολύ προσωπικό. Είπατε ότι όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πακέτο με τα υπόλοιπα μέσα. Αυτό δεν εξαρτάται τόσο από μένα. Αυτά θα συζητηθούν και στην ομάδα ο Μάουρο εδώ είναι, εδώ ο κύριος Μπροκ, ο κύριος Λάμστορφ θα συμμετέχουν. Και θα δούμε τι θα προκύψει και από την ομάδα λοιπόν. Νομίζω ότι ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα καταλήξουμε σε μια σωστή λύση Άρα προσβλέπω στις διαπραγματεύσεις αυτές και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα οριστικοποιηθεί ακόμα η πρόταση γιατί κινούμαστε παράλληλα και με τα υπόλοιπα μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω εκ νέου. Αν υπομονώ να δω και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Grazie. Qualche momento di pausa. Ένα διάλειμμα. Περιμένουμε τους εισηγητές για το επόμενο σημείο. Ευχαριστώ. Διάλειμμα. Επόμενο σημείο. Σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας με τη Ρωσία. Πάμε στην παρουσίαση της μελέτης «Πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη Ρωσία το 2012» κατόπιν του νέου ρόλου της Ρωσίας στο διεθνές κοινικό ανατέθηκε μία μελέτη στις τωρινές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα το ρόλο της Ρωσίας στο, στο διεθνές σενάριο. Ε, ο παράγοντας που είχαμε είναι οι πρόσφατες εκλογές, οι διαπραγματεύσεις νέας, της νέας συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, προσχώρηση της Ρωσίας στην ΠΟΕΦ, και επίσης γεωπολιτικές περιοχές που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη Ρωσία, Βόρεια Κορέα και Συρία. Θέλουμε να αξιολογήσουμε την ε, δυνατή εξέλιξη της, ε, της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, εξέλιξη της οικονομίας, εμπλοκή των σχέσεων Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και προοπτικές διαπραγμάτευσης της νέας συμφωνίας Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία ο καθηγητής Φίλψον του Chat Mouse για 10 λεπτά να μας παρουσιάσει. Chatham House, συγγνώμη. Η έκθεση αυτή συνεγράφει από ένα οικονομολόγο και ένα πολιτιολόγο και εγώ είμαι ο οικονομολόγος σήμερα, οπότε θα πρέπει να δείξετε κάποια ανοχή μαζί μου. Το κύριο ερώτημα είναι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα μια πιο ανοιχτή Ρωσία και εγώ θα βασιστώ περισσότερο στο οικονομικό κομμάτι αυτής της ερώτησης. Έχω κάποιο σκεπτικισμό για αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Ίσως δεν θα δούμε τόσο μεγάλες αλλαγές στη Ρωσία όπως υποστηρίζουν οι ορισμένοι, αλλά ας δούμε πρώτα ποια είναι τα θέματα. Πρώτα απ' όλα, η Ρωσία αντιμετωπίζει ένα σύνολο από προκλήσεις για το άμεσο μέλλον, που είναι και μια ευκαιρία να γίνει πιο ανοιχτή προς τον έξω κόσμο. Περιμένουμε και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί όλα αυτά δεν έχουν κυρωθεί ακόμα από το Ρωσικό Κοινοβούλιο. Περιμένουμε να υπάρξει προσχώρηση στον ΠΟΕ από τη Ρωσία στο τέλος του καλοκαιριού. Αλλά υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία επίκυνται που θα έχουν και εκεί δυνατότητες για ένα πιο ανοιχτό πνεύμα, η Προεδρία των G20 από τις αρχές Ιουλίου, η διάσκεψη κορυφής ε, για τη συνεργασία ε, με την, Ασία, που θα γίνει στο Βλαντιβοστόκ με οικοδεσπότη τη Ρωσία. Πάλι υπάρχουν δυνατότητες ότι θα γίνει μέλος της ΟΣΑ, του ΟΣΑ, η Ρωσία του χρόνου. Η Ολυμπιακή στο Σότσι, η χειμενή Ολυμπιακή το 2014 στο Σότσι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2018 Είναι λοιπόν ευκαιρίες που η Ρωσία θα ανοίξει τις πόρτες της στον έξω κόσμο. Ε, αυτά τα οποία θα προκύψουν από το ΠΟΕ είναι σαφή, δεν θα έχουμε δασμούς, θα υπάρχουν όρια για τις αγροτικές επιδοτήσεις, τεχνική έλεγχη στα σύνορα και στα τελωνία όπως έχουν γίνει δεκτοί σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή άρση των υπερβολικών περιοριστικών προστατευτικών ε, μέσων, άνοιγμα για τις διεθνείς επενδύσεις, καλύτερη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Μέτρα που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις και το εμπόριο, όπως πραγματικά το να ζητά κανείς τοπικό περιεχόμενο στα συναρμολογούμενα αυτοκίνητα και τα λοιπά, όλα αυτά πρέπει να έρθουν. Τώρα δεν θα γίνουν αυτά αμέσως. Κάποια από αυτές τις δεσμεύσεις θα πρέπει να εγκριθούν αμέσως με την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Κάποια άλλα όμως θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. 40% των δασμών θα πρέπει να τροποποιηθούν αμέσως και άλλα κομμάτια σε τρία χρόνια. Οι επιδοτήσεις για το μέταλλο σκράπ θα μειωθούν στο μέλλον και τα λοιπά. Αλλά κάποιες από τις προσαρμογές που έχει διαπραγματευτεί μέχρι στιγμής η Ρωσία είναι κατά την άποψή μου αρκετά γενναιόδορες για τα συμφέροντα της Ρωσίας. Χρειάστηκε να υπάρξουν λοιπόν πολλές παραχωρήσεις για, από την πλευρά πολλών χωρών, πάνω από 15 χώρες έχουν δείξει ενδιαφέρον για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό της προσχώρησης της Ρωσίας. Εκεί που είναι το σημαντικό θέμα είναι πώς θα γίνει η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Η προσχώρηση στον ΠΟΕ κάνει μια χώρα να είναι υπόλογη σε διεθνές επίπεδο. Αλλά οι μηχανισμοί αυτή επίλυσης διαφορών στον ΠΟΕ δεν λειτουργούν με ταχύτητα, δεν καταλήγουν σε μια ικανοποιητική και γρήγορη επίλυση των διαφορών. Πολλοί από σας γνωρίζετε τις μακροχρόνιες διαμάχες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τη διαμάχη Boeing-Airbus σε σχέση με τις επιδοτήσεις από τις δύο πλευράς. Αυτά μπορούν να κρατήσουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ θα έλεγα ότι η κύρια πίεση για τη μεταρρύθμιση στην οικονομία της Ρωσίας δεν είναι οι προκλήσεις αυτές όπως η προσχώρηση στον ΠΟΕ. Αυτό το οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο είναι τα θέματα της ε, αντιμετώπισης των χαμηλών τιμών πετρελαίου που θα είναι το κυριότερο κίνητρο για την μεταρρύθμιση. Χρειάζεται μια μεταρρύθμιση όπως αναφέρουμε και στην εκθεσή μας. Και στις οθόνες παρουσιάζουμε και τη βαθμολογία της, Ευρω... της Ρωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι από 183 χώρες σε, στην 120η θέση συνολικά. Οι καλύτερε τώρα εκτιμήσεις που έχουμε και είναι <clears throat> αισιόδοξε για τα αποτελέσματα σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα της Ρωσίας σε επίπεδο ΑΕΠ, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο μέχρι το 2020, είναι περίπου 3,3% μεγέθυνση του ΑΕΠ σε αιτήσιο επίπεδο. Εδώ σας δείχνω το άνω όριο, ένα πιστευτό αν και ε, αισιόδοξο επίπεδο μεγέθυνση 5%. Η πιο κάτω γραμμή είναι η γραμμή του 2,5% ετήσια μεγέθυνση και αυτά δείχνουν τα πιθανά σενάρια και το αποτέλεσμα του, της προσχώρησης στον ΠΟΕ θα μας δώσει το 3,3% που ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν τα σενάρια τα οποία είναι τα πιο αισιόδοξα και τα πιο απεσιόδοξα. Η προσχώρηση στον ΠΟΕ θα οδηγήσει πράγματι και σε βελτιώσεις στην οικονομική ελευθερία. Έχουμε μέτρα που έχουμε με δείκτες για την οικονομική ελευθερία σε πολλές χώρες. Έχουμε χώρες που ήταν στο παρελθόν κομμουνιστικές, η Αρμενία, η... η Αρμενία λοιπόν, η Κίνα, η Γεωργία και η Ουκρανία. Η Κίνα δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα. Η Ουκρανία όχι, η Αρμενία λίγο και η Γεωργία έχει βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ελευθερία, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι απαραίτητα η προσχώρηση στον ΠΟΕ μια επιρροή προς την κατεύθυνση αυτή. Το status quo στη Ρωσία. Βλέπουμε την μπλε γραμμή εδώ. Έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη ευμάρεια στη Ρωσία. Ιδιαίτερα την εποχή 2008 2009 μέχρι την εποχή 2008-2009 που χτύπησε η κρίση. Μετά όμως ξανά ήρθε η ανάπτυξη. Έχουμε την άλλη γραμμή, το, τη ρόζη, η οποία είναι η κατανάλωση των οικοκυριών και η κάτω γραμμή δείχνει την ένδια, η οποία αυξάνεται, η οποία μειώνεται μάλλον. Ένα από τα θέματα τα οποία θέσαμε είναι αν θα υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα από την ε, προσχώρηση των ΠΟΕ σε σχέση με τις περιφερειακές ανισομέρειες. Η καλύτερη λοιπόν εκτίμησή μας είναι, είναι ότι λόγω της προσέλκυσης ε, επενδύσεων θα υπάρξει μια μεγάλη βελτίωση στην Άπο και στην βορειοδυτική ε, Ρωσία. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι η περιοχή της Μόσχας θα εξακολουθήσει να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη. Εδώ όμως βλέπουμε και το ποσοστό ανεργία σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Αυτό δείχνει και κάποια στοιχεία που είναι εντυπωσιακά. Κάτω από 2% ανεργία στη, Μωσία στη Μόσχα, 49,7% στην Οικουσετία, δίπλα στην Τσετσενία, 50% σχεδίων. Και η διακυμάνσεις είναι τεράστιες μεταξύ των διαφόρων αυτών περιοχών. Τιμές πετρελαίου και ΑΕΠ έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Έχουμε δύο κλίμακες, μιλάμε όμως για τα ίδια ποσοστά. Η κόκκινη γραμμή δείχνει την ε, κίνηση του ΑΕΠ, η μπλε γραμμή δείχνει τις τιμές του πετρελαίου από τα ουράλια. Κάνουμε μια ε, προεκβολή μέχρι το 2020 και οι ρωσικές προβλέψεις με κάπως αισιόδοξο τρόπο θεωρούν ότι θα υπάρξει μια σταθεροποίηση, μια μικρή αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Αλλά η τιμή του πετρελαίου έχει κινηθεί με πολύ μεγάλη δοκιμάσει στο παρελθόν και μάλλον θα συνεχίσει να το κάνει. Συμπεράσματα. οι προσχώσει στον ΠΟΕ θα βοηθήσει δυνητικά σε περαιτέρω φιλελευθερωποίηση τη ρωσική οικονομία και κοινωνία. Υπάρχουν όμω πιο σημαντικέ επιρροέ και επιδράσεις για την κοινωνία και την οικονομία τη Ρωσία για την μεταρρύθμιση που θα προκύπτουν περισσότερο από εγχώριες πιέσεις, οι διαδηλώσεις, κινητοποίησεις στους δρόμους εξακολουθούν να συνεχίζονται. Δεν είναι καθόλου σαφές τι θα γίνει με τη νέα κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε πολύ καλά ακόμα ποιος θα είναι μέσα. Έχουμε απλώς φήμες και φημολογία. Μόνο στις 15 του μηνός θα γνωρίζουμε καλύτερα. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι οι τιμές του πετρελαίου. Ακόμα και αν γίνει η προσχώρηση στον ΠΟΕ και η Ρωσία αναλάβει τις υποχρεώσεις της και τις εφαρμόσει πλήρως, το, η επιρροή του, της προσχώρησης δεν είναι επαρκής για να αλλάξει πολύ τα πράγματα. Απλώ μπορεί να υπάρξει μια συνέργεια μεταξύ μεγαλύτερης ανοιχτή στάση προς τον έξω κόσμο και εγχωρίων πιέσεων. Αλλά δεν μιλάμε για μεγάλη μετατόπιση στις οικονομικές προοπτικές της Ρωσίας που να οφείλονται μόνο στην προσχώρηση στον ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η δεύτερη τοποθέτηση είναι ο κύριος Χόμποντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω δύο λόγια στα αγγλικά. Συμφωνώ με τα συμπεράσματα, απόλυτα. Όντως, ο ΠΟΕ δεν αλλάζει πάρα πολλά στις δομές και στις ιδιομορφίες της Ρωσίας. Αυτό ισχύει και για άλλες χώρες. Από την εμπειρία μας με άλλες χώρες, όπως η Κίνα, προκύπτει ότι για μεγάλες ε, χώρες όπου δεν αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά υπάρχει πιο ανοιχτός χαρακτήρας, πιο πολλής ανταγωνισμός και μπορεί να περιοριστεί η εξουσία κάποιων μεγάλων ε, ομίλων, κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μάλλον και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πιο σωστή αντιμετώπιση, πιο δίκαιη αντιμετώπιση αν συνδυαστεί η προσχώρηση στον ΠΟΕ με κάποιες νομικές βεβαιότητες, αυτό είναι πιο σημαντικό για μας, νομικές βεβαιότητες για τους επενδυτές και με μείωση της διαφθοράς. Αν λοιπόν σε σχέση με τα στοιχεία αυτό προωθηθούν και οι διαστάσεις αυτές, η προσχώρηση στον ΠΟΕ θα έχει θετικό αντικτύπο στην διαδικασία εξχρονισμού της Ρωσίας για την τιμή του πετρελαίου. Και πάλι η υψηλή τιμή του πετρελαίου περιορίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις. Αν ήταν πιο χαμηλή η τιμή του πετρελαίου θα υπήρχε πιο μεγάλη πίεση για μεταρρυθμίσεις. Αλλά αναμένω ότι θα παραμείνει υψηλή η τιμή του πετρελαίου γιατί η παγκόσμια οικονομία θα ξαναξεκινήσει να αναπτύσσεται και άρα η τιμή του πετρελαίου θα παραμείνει υψηλή. Αυτό θα περιορίσει λοιπόν την ε, ανάγκη, την πιεστικότητα διεξαγωγής ε, μεταρρυθμίσεων και ακόμα και κάποιες δεσμεύσεις που έχουν αναλευθεί από τον ε, Πούτιν. Αν προκύψει τώρα παγκόσμια ύφεση, μπορεί να πέσει κάπως η τιμή του πετρελαίου και έτσι θα πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στη Ρωσία δεν σημαίνει αυτό φυσικά ότι θέλω να υπάρξει ύφεση για να, παγκόσμια για να υπάρξει τέτοια πίεση στη Ρωσία. Τρίτον, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, γιατί αυτό δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στον οικονομικό κλάδο, στον ακαδημαϊκό κόσμο, στα πανεπιστήμια, αν υπάρξει και κάποια απελευθέρωση στο καθεστώς στη Ρωσία για να εισέλθουν πιο πολλοί αλλοδαποί στη Ρωσία. Αυτό χρειάζεται νομίζω στην Ρωσία. Πιο πολύ επαφή, πιο πολύ ανεκτός χαρακτήρα με τις δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και αυτό στη μέση τάξη, γιατί φυσικά η υψηλές ε, μισθολογικέ ε, τάξεις ε, έχουν επαφές με την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό όμως που χρειάζεται. Η μέση τάξη έχει δυσκολία να λάβει θεώρηση και εδώ θα βοηθούσε η απελευθέρωση. Επίσης θα βοηθούσε μια πιο ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Βλέπουμε ότι παρεκκλίνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από τις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί και η Ουγγαρία με τον Αμπόκο, για, παράδειγμα, κάνει πιο πολλές χάρες στη Ρωσία και άλλες χώρες, μην, δεν είναι μόνο η Ουγγαρία. Αυτό είναι πρόβλημα. Αν ήταν πιο ε, ενωμένη η στάση μας, έναντι της Ρωσίας θα είχαμε πιο μεγάλο αντίκτυπο. Και αυτό ασφαλώς περιλαμβάνει και καταστάσεις, ε, τη δύσκολη κατάσταση με την Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για την τελεωνική ένωση μεταξύ Ρωσίας, Καζακστάν και Ουκρανίας. Συνολικά νομίζω ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να διαδραματίζει τέτοιο ρόλο εξισορροπητικό μεταξύ συμφωνίας με την Ανατολή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ήμουν κι εγώ πολιτικός στη Ρωσία το ίδιο θα έκανα. Θα προσπαθούσα να εξισορροπήσω τους διαφόρους τομείς για να συνδυάσω όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι από ευρωπαϊκής πλευράς θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση για τα θέματα αυτά. Να είναι πιο ισχυρή η κοινή μας θέση, γιατί ασφαλώς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντιδράσει και πιο ηχηρά η Ρωσία στις δικές μας θέσεις. Άρα, συνολικά, στο θέμα των διαπραγματεύσεων ε, και τις συμφωνίες ε, PCA μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος αν υπάρξει κάποια συμφωνία στο θέμα των θεωρήσεων, νομίζω ότι θα σημειωθεί κάποια παραπάνω πρόοδος για το θέμα της ενέργειας. Λυπάμαι που είμαστε ακόμα κατακαιρματισμένοι σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας με στη Ρωσία. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το ενδιάμεσο καθεστώς θα παραμείνουν οι σχέσεις μας με τη Ρωσία. Θα δούμε τι θα προκύψει και από τη νέα κυβέρνηση που θα πρέπει να σχηματιστεί τις επόμενες ημέρες. Αν μείνουμε σε αυτή την κατάσταση απολυταρχικής πολιτικής που κάνει μεν υπαναχωρήσεις αλλά δεν αλλάζει στη δομή της, λυπάμαι επίσης γιατί φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένη η κοινωνία των πολιτών μετά τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες πραγματικά πρέπει να πω ότι τις βλέπω με επικριτικό πνεύμα. Δεν είναι πραγματικές μεταρρυθμίσεις, δεν είναι πραγματικός τρόπος να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Δεν βλέπω στην παρούσα φάση να υπάρχουν οι όροι, οι συνθήκες για μια μεγάλη πρόοδο. Ίσως σε κάποιους τομείς να σημειωθεί πρόοδος, σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, πολιτικών που θα προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν την διαφθορά, θα προσπαθήσουν να προωθήσουν τα συμφέροντα των δήμων του, εκεί θα υπάρχει πραγματικά συμφέρον προκειμένου να δώσουμε βοήθεια σε αυτούς τους κυβερνήτες. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πραγματιστές στην προσέγγισή μας, αλλά να επικρίνουμε σε περιπτώσεις ε, παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων και να παρακολουθούμε και το θέμα του ΠΟΕ. Αν προσχωρήσει τον ΠΟΕ, το οποίο είναι θετικό, να εφαρμόσει αυστηρά τους σχετικούς όρους, γιατί στην Ρωσία το κράτος δικαίου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, όχι μόνο για την κοινωνία των πολιτών, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κνούτ Φλέκεστάιν, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της ε, μειχτής αντιπροσωπείας. Μεγάλος ο τίτλος, αλλά σύντομος ο λόγος. Στα γερμανικά. Ο κύριος ε, Σφόμποντα αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της μελέτης. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε γιατί δεν έχω διαφωνία με αυτά που λέει, απλώς όμως δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Το λέω αυτό θετικά. Δεν σημαίνει ότι είναι δυσνόητη η έκθεση. Λέει ότι μπορεί να βοηθήσει η προσχώρηση στον ΠΟΕ, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Αλλά είναι άλλα πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν περισσότερο την κατάσταση. Όσοι εκεί κατάλαβα. Θα περιοριστώ σε δύο ερωτήματα μονάχα. Το πρώτο ερώτημα αφορά τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας για μια συμφωνία συνεργασίας. Πολλοί εκπρόσωποι της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και πολλοί εκπρόσωποι των επιχειρήσεων της Ευρώπης στη Ρωσία έχουν δώσει την εντύπωση ότι η προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα μπορούσε να είχε μια θετική επίδραση στις βραδιπορούσες αυτές διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία με τη Ρωσία. Τώρα είναι ασαφής ίσως η μελέτη και ίσως ελαφρά αισιόδοξη. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε προβλήματα με την έλλειψη συμφωνίας για τα θέματα ενέργειας και υπάρχουν και άλλοι λόγοι επίσης οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Το ερώτημά μου λοιπόν θα ήταν σε εσάς Ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ενδεχόμενη συμμετοχή τη Ρωσία στον ΩΣΑ, κάτι το οποίο το διαλαμβάνει επίση και η εκθέσή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στον, στον κύριο Βίλαντ και στον κύριο Κυρίλοφ. Την κυρία Όιλαντ, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα το όνομά μου. Συγγνώμη, ήταν κακή προφορά, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και την έκθεση που έχετε παρουσιάσει, η οποία φαίνεται να είναι εμπεριστατωμένη και πλήρως και εστιάζει πάρα πολύ στο ΠΟΕ και την προσχώρηση της Ρωσίας. Φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα για τη Ρωσία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια θα μπορέσει να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες για το εμπόριο. Το ερώτημά μου όμως είναι και αυτό το οποίο θα ήθελα να ακούσω από τα χείλη του εμπειρογνώμου που μας παρουσίασε αυτή την έκθεση πώς εκτιμάτε τα θέματα της διαφθοράς εκεί. Αναφερθήκατε το, στο θέμα της διαφθοράς στη Ρωσία, αλλά εγώ διάβασα πρόσφατα στη μία έκθεση του, της εξαμνής σκέψης Ίντεμ ότι εκτιμούν ότι 35% της ρωσικής οικονομίας χάνεται στη διαφθορά. Δεν χάνονται μονάχα σε τοπικό επίπεδο, είναι πολλές φορές και σε κεντρικό επίπεδο πολιτικής ηγεσία όπου φτάνει αυτή η διαφθορά. Θα ήθελα να έχω λοιπόν κάποιες ε, ιδέες από εσά για το πώς η προσχώρηση στον ΠΟΕ αν θα, μάλλον, κατά πώς θα αλλάξει την κατάσταση αυτή και αν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση αυτή και το διεφθαρμένο αυτό σύστημα. Και η δεύτερη τώρα παρατήρησή μου, για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στη Ρωσία πρέπει να δούμε τις για στο επιχειρηματικό κλίμα. Εδώ υπάρχει από μια πλευρά το πρόβλημα τη διαφθοράς, από την άλλη πλευρά υπάρχει η έλλειψη κράτους νόμου και δικαίου. Και εδώ θα αλλάξει αυτό με τη συμμετοχή στον ΠΟΕ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανονισμών σε εσωτερικό επίπεδο για την ε, εφαρμογή και στο εσωτερικό της Ρωσίας του ΠΟΕ. Γιατί μέχρι στιγμής από την πλευρά της Ρωσίας Έχουμε δει τόσα πολλά προβλήματα σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, ιδίω για τι επιχειρήσει. Ο Κυριλόφ. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξής. Την ανάλυση αυτή που βασικά τις οικονομικές ε, πτυχές ε, δεν ακούσαμε τίποτε για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας. Υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι θα, υπήρξε, θα υπήρχαν διασυνοριακές επενδύσεις, κοινά project και το καθεξής. Ουσιαστικά όμως τίποτα δεν έχει πραγματοποιηθεί σε ό,τι αφορά το ανατολικό τμήμα αυτό της Ρωσίας. Πρόσφατα, για πρώτη φορά, υπήρξε ένα κρίσιμο άρθρο, στη, μάλλον επικριτικό άρθρο στην Κίνα για τον τρόπο ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας. Όλα αυτά συνδέονται, αλλά επειδή αναφέραμε την Κίνα, εγώ πιστεύω ότι συμφέρει τη Ρωσία να επιλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ουτέρο. Σε ό,τι αφορά την Κίνα δηλαδή, η Ρωσία χρειάζεται την Ευρώπη και αντίστροφα. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά τα εμπόδια της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, αλλά υπάρχει και άλλη μία πτυχή σε όλα αυτά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στη Ρωσία προβάλλεται κυρίως η μέση τάξη. Σε ό,τι αφορά την οικονομική ελευθερία, Κυρίως ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που πλήττονται και υποφέρουν από την κατάσταση αυτή. Χωρίς την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νομίζω ότι η ρωσική οικονομία ασφαλώς θα βρίσκεται σε μια βαθιά ύφεση για μακρόχρονικό διάστημα και κατά δεύτερον συμφωνώ με το ε, δυνητικό αποτέλεσμα, αντίκτυπο της απελευθέρωσης από το καθεστώς της ε, βίζας των θεωρήσεων. σε ό,τι αφορά ό,τι την, την αντιπυραυλική άμυνα τώρα, θα ήθελα να θέσω και αυτό το θέμα και να μου πείτε τι γίνεται. Ο κύριος Σούλς έχει το λόγο. Μία ερώτηση προς τον κύριο Χάνζεν Τι μας κάνει να ελπίζουμε ότι με την προσχώρηση στον ΠΟΕ η Ρωσία θα βελτιώσει την νομική βεβαιότητα που επικρατεί στην επικράτειά της. Δεν είναι ε, και είναι γνωστό αυτό κράτος δικαίου. Ακόμα και ο πρώην πρόεδρος Μετβέντεφ ε, κατέγγειλε τον... Ε, Πρέπει να πούμε όμως ότι δεν σημειώθηκε προβελτίωση ε, στην διαφθορά και στην καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολουθεί να αποτελεί συστατικό της Ρωσίας ε, η διαφθορά. Άρα σε τι ελπίζουμε, σε τι στηρίζουμε τις ελπίδες μας ότι θα περιοριστούν τα προβλήματα αυτά λόγω της προσκόρησης των ΠΟΕ. Ο κύριος Σβόμποντα δεν διαπράττουμε σφάλμα αν ε, εξισώνουμε την ελευθερία ε, ταξιδίων με την ελευθερία ε, θεωρήσεων. Έχει ελευθερία για ταξίδια η Ρωσία. Δεν θα ήταν σημαντικότερο να επισημάνουμε ότι στη Ρωσία υπάρχει έλλειμμα, ακραίο έλλειμμα σε άλλες ελευθερίες, όπως η ελευθερία του διαδηλώνει. Είδαμε στις 6 Μαΐου πώς ε, περιορίζονται οι ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συναθρίζεσαι, ε, της ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των θεωρήσεων ε, δεν είναι το πιο κατεπήγον ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ρωσία σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε, στις επιδράσεις της τιμής του πετρελαίου. Δεν συμφωνώ. Ότι τα πράγματα έχουν όπως παρουσιάζεται στην ε, έκθεση που λέει ότι αν συνεχιστούν οι υψηλές τιμές ε, πετρελαίου θα εμποδίσουν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης και η πτώση της τιμής πετρελαίου θα ευνοήσει τις αιτήσει μεταρρύθμισης. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα. <clears throat> Πάρτε το παράδειγμα της Κίνας. Όπου η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον φαίνει κάτι περισσότερο αλλά στην περίπτωση της Ρωσίας η κατάρρευση της ε, τιμής του πετρελαίου δεν δίνει ένα αίσθημα κατεπήγοντας. Απλώς αυξάνει την ε, εξουσία των εξτρεμιστών <clears throat> γιατί οι μέσες τάξεις χάνουν την ελπίδα τους. Που να αυξήσει τη δυνατότητα φασισμού. Έτσι λένε πολλοί από τους εμπειρογνώμονες, ιδίως στην Φιλανδία. ότι η κατάρρευση του επίπεδου διαβίωσης στη Ρωσία μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες. και δεν θα αυξήσει την ε, αίτηση για μεταρρυθμίσει, μάλλον το αντίθετο. Ο κύριος Μίλαν Μόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα δύο ερωτήσεις. Τι ελπίζουν από τη Ρωσία ως επόμενη Προεδρία του G20 Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ρωσίας σε αυτό το φόρουμ. Δεύτερο, πώς θεωρείτε ότι εκτιμάει η Ρωσία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν της, ε, δεν της έδινε και πολλή αξία στο παρελθόν. Πάντοτε ευνοούσε περισσότερο τις διμερείς συμφωνίες με τις ε, μεγάλες χώρες. Τώρα σήμερα με το χρέος και την κρίση. Ποια είναι η στάση της Ρωσίας, ο κύριος Σούεφλιντ; Σας ευχαριστώ κύριε <clears throat> Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Φιλ Χάνσεν. Δύο ερωτήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Πώς η δημογραφική κάμψη επηρεάζει την αγορά εργασίας με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και κατά πόσο θεωρείτε ότι η κάμψη αυτή στην αγορά εργασίας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη μετανάστευση προς τη Ρωσία με αντίστοιχα προβλήματα. Ολοκληρώσαμε με τους ομιλητές, παρακαλώ. Έχετε το λόγο για τις απαντήσεις. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την πολυπληθώρα ερωτήσεων. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω επιτυχώς σε όλες αυτές. Πολλές από αυτές είχαν να κάνουν με το θέμα της, ε, του κράτους δικαίου ή της απουσίας και της αδυναμίας του κράτους δικαίου στη Ρωσία. Και το ερώτημα ήταν γιατί η προσχώρηση στον ΠΟΕ θα μπορούσε να επηρεάσει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι βλέπουμε ότι η Κίνα η οποία έγινε μέλος του ΠΟΕ εξακολουθεί να έχει μια σχετικά ολέθρια πόλη, απουσία κράτους δικαίου. Δεν υπάρχουν λοιπόν εγγύησεις, δεν υπάρχουν βεβαιότητες για το θέμα αυτό. Η ελπίδα μας τώρα είναι ότι η ανάγκη να υπάρξουν να υπάρξει συμμόρφωση με τεχνικά, τεχνικές προδιαγραφές και φυτο-υγειονομικά πρότυπα είναι πολύ θετικά. Όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να φαίνονται μικρά και κούτσικα σε λεπτομέρεια απαιτούν από την Ρωσία να απαντήσει και στις ερωτήσεις και τις αιτιάσεις των εταίρων της. Κάποιος που είναι στον ΠΟΕ δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Το να δεχτεί λοιπόν διεθνή πρότυπα ή τουλάχιστον το να προσπαθήσει να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα θα έχει θετικό αποτέλεσμα η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δύσκολο. Η ιδέα της Ρωσίας για την της εξουσίας στη Ρωσία θεωρούν ότι μια παράξενη οργάνωση που δίνει τόσο πολύ εξουσία σε μικρές χώρες. Η Ρωσία σκέφτεται με όρους μεγάλων δυνάμεων, περιφερειακών δυνάμεων. Η ρωσική ελίτ θέλει να αντιμετωπίσει αυτές τις περιφερειακές δυνάμεις που θεωρεί ότι είναι σημαντικές. Δεν θέλει να ασχολείται με μικρότερες δυνάμεις. Δεν κατανοούν λοιπόν πολύ καλά τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος. Κατά πόσο το επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να είναι η προσχώρηση στον ο ΩΣΑ θα δώσει περισσότερη δύναμη πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω. Ένα από τα στοιχεία είναι ότι το να προσπαθήσει να μπει η Ρωσία στον ΠΟΕ, η διαδικασία αυτή κάνει τη, στην Ευρωπαϊκή, δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια όπλα. Να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο των προτύπων της Ρωσίας. Όταν γίνει μέλος της, ε, του ΩΣΑ η Ρωσία, που μπορεί να μην πολύ γρήγορα, τότε ενδεχομένως θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση προς τη Ρωσία σε σχέση με την οικονομία της αγοράς και τον ανταγωνισμό στην αγορά. Ο έχει ασκήσει πίεση σε σχέση με τέτοιου είδους θέματα. Εγώ ήμουνα παρόν στις διάφορες ε, παρακολουθήσεις που έχει γίνει με τη Ρωσία για τα θέματα αυτά και όταν μιλάει κανείς με τους Ρώσους υπεύθυνους, μιλά την ίδια γλώσσα με σένα. Αλλά όταν δούμε την έκθεση των Ρώσων για, ε, ε, τα μέτρα που έγιναν σε σχέση με τη στρατηγική του 2020 εκεί, όλοι μιλάνε για την ανάγκη να υπάρξει ισόπεδο γήπεδο ανταγωνισμού, ανεξάρτητη δικαστική εξουσία. Είναι όλα αυτά η κλασική φιλελεύθερη επιχειρηματολογία. Όλοι αυτοί που δεν είναι μέσα στα κέντρα εξουσία μιλάνε για το θέμα αυτό, ακόμα και κάποιοι φιλελεύθεροι μέσα στα κέντρα εξουσία. Αλλά αυτό το οποίο δεν λένε είναι πώ θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο στην πράξη. Θα παραλείψω μερικά θέματα που αναφέρατε, αλλά να σταθώ στο θέμα της δημογραφικής αλλαγής. Ξέρουμε ότι ο συνολικός πληθυσμός της Ρωσίας έχει μια πτωτική τάση Υπήρξαν κάποιες διορθώσεις στην τελευταία απογραφή, αλλά πρόσφατα είναι φανερό ότι μειώνεται και ο αριθμός του ενεργού εργασιακά πληθυσμού και το λέει και η έκθεση. Και οι προ... προβλέψεις της στατιστικής οργάνωσης Ρωσίας για τον πληθυσμό, που, για τον ενεργό πληθυσμό που περιλαμβάνουν τους, ακόμα και τους μετανάστες μέχρι το 2020 είναι μία μείωση η οποία πλησιάζει και μία μείωση που μπορεί να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια μεταξύ του 2010 και 2020. Αυτό είναι ένας από του κύριου λόγου για τους οποίους μπορούμε να περιμένουμε ότι οι λήπτες αποφάσεων στη Ρωσία μπορεί να χρειαστεί να πιέσουν περισσότερο για βελτίωση της παραγωγικότητας. Υπάρχουν λοιπόν κίνητρα για αλλαγές και το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί αυτό που θέλουν οι Ρώσοι είναι μετανάστες με καλύτερα προσόντα όπως και οι περισσότερες χώρες στον κόσμο. Αυτοί όμως που έρχονται είναι κυρίως <clears throat> ανειδίκευτοι, κυρίως από τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Και αυτό οδηγεί βέβαια σε κοινωνικές εντάσεις. Υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν. Ο πρόεδρος Βόμποντα. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ερώτημα του κυρίου Σούλτς. Εγώ δεν αναφέρθηκα στο θέμα της ελευθερίας ταξιδίου στα θέματα των ελευθεριών. Απλώς αναφέρθηκα στο θέμα τι μεγαλύτερε ελευθερίες στο εσωτερικό της Ρωσίας και τις μεγαλύτερε ελευθερίες για την ε, μέση τάξη στη Ρωσία. Δεν αναφέρθηκα στα θέματα διευκολύνσεων βίζα, λοιπόν. Για τις επαφές όμως είναι απαραίτητο όλο και περισσότερο να δώσουμε μια υποστήριξη στα στρώματα της μέσης τάξης στη Ρωσία. Έχουμε δει στα διάφορα προγράμματα ότι αυτά είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολύ σημαντική η επαφή ιδίω για τα κινήματα της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, στους οποίους θα πρέπει να παρέχουμε και την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Επόμενο σημείο. Έκθεση του κυρίου Σαΐντ Αλχαντράουι των πεπραγμένων ε, στην αποστολή στο Μασρέκ ε, από τις 30 Απριλίου στις 4 Μαΐου του 2012. Επίσης ένας απεσταλμένος της αντιπροσωπείας πήγε στην Αίγυπτο, είχε και επαφές με τις Αιγυπτιακές αρχές και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και του, και του κλήρου. Παρακαλώ τον συνάδελφο να μας περιγράψει την επίσκεψη, να μας πει τη γνώμη του και να μας αναφέρει πώς έχει κατάσταση στην Αίγυπτο. Οικονομία και ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο για να σας αναφέρω για την επίσκεψή μας την προηγούμενη εβδομάδα είναι η πρώτη ε, μειχτή αντιπροσωπεία μετά τις εκλογές. και που άλλαξαν τη μορφή. Ε, λοιπόν, ας αφήσουμε τον εισηγητή να εκφράζεται όπως νομίζει. Έλεγα λοιπόν ότι το κοινοβούλιο άλλαξε όψη, διότι Σήμερα επικρατούν οι Ισλαμιστές δύο τάσεων. Έχουμε το πολιτικό σκέλος των αδερφών μουσουλμάνων και το πολιτικό κόμμα Αλμούρ. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα ορίστηκε από σφραγίστηκε μάλλον από την βούληση του στρατού. Και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς στο μέλλον θα εξελιχθούν οι καταστάσεις και οι σχέσεις μεταξύ νομοθετικού και εκτελεστικού νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Πρόκειται για ένα πολιτικό χάος με συνεχείς ε, συγκρούσεις τον τελευταίο καιρό μεταξύ της Ισλαμικής πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου και από την άλλη των στρατιωτικών αρχών που εξήγηλαν ότι θέλουν ότι θα, να ότι θα αφήσουν την εξουσία μόλις εκλεγεί ένας νέος πρόεδρος. Τώρα το Μάιο θα έχουμε τον πρώτο γύρο των εκλογών, των προεδρικών εκλογών. Και παράλληλα γίνεται και η συζήτηση για το νέο σύνταγμα. Δεν ξέρουμε εάν το σύνταγμα θα εγκριθεί πριν ή μετά τις εκλογές. Είναι πολύ πιθανό να εγκριθεί μετά τις εκλογές. αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να εκλέξουν οι Αιγύπτιοι έναν πρόεδρο χωρίς να ξέρουν τι εξουσίες θα έχει. Με λίγη διαφάνεια δηλαδή. Έχει δημοσιευθεί από την Εκλογική Επιτροπή ο κατάλογος των υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές. Δημιουργήθηκαν και ιστορίες με την επιλογή διότι ο υποψήφιος της αλαφικής ε, τάσης ε, αποκλείστηκε. Έγιναν διαδηλώσεις, συγκρούσεις, στο Υπουργείο Αμήνης παρενέβηκε ο στρατός και δύο μέρες μετά Είχαμε άλλες συγκρούσεις με 11 νεκρούς και την προηγούμενη εβδομάδα την Παρασκευή είχαμε διάφορες διαδηλώσεις στο Κάιρο. Χαοτική κατάσταση. Οι συμμαχίες αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν είναι καθόλου ιδεολογικές. Ο Αμπτούλ Φουτού μαζί με τον Αντερμούς είναι τα φαβορή για τις προεδρικές εκλογές. Ο δε πρώτος αποχώρησε από τους αδερφούς μουσουλμάνους γιατί θα ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του Και αυτό το έκανα όταν οι αδερφοί μουσουλμάνοι δήλωσαν ότι δεν θα παρουσίαζαν υποψήφιο. Και αποχώρησε για να γίνει υποψήφιος και τον υποστηρίζει τώρα ένα κρέος αλαφικό κόμμα. Όπως επίσης και ο περίφημος blogger τον οποίο είχαμε υποστηρίξει και εμείς στο παρελθόν, υποστηρίζει τον Αμάρτ Έχουμε λοιπόν έναν υποψήφιο ο οποίος είναι λιγότερο χαρισματικός. Μιλάμε για προεδρικές εκλογές λοιπόν σε δύο γύρους, άρα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν πολλές πολιτικές συζητήσεις. Και τους τελευταίους μήνες το Κοινοβούλιο έχει καταστεί όλο και λιγότερο δημοφιλές. Οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις προβληθήκαν και στην τηλεόραση και έτσι το ευρύ κοινό παρακολουθεί το τι συμβαίνει με ιδιαίτερη διαφάνεια. Αλλά καταλήξαμε στην διαπίστωση ότι μεγάλο τμήμα της συζήτησης ε, δεν έχει να κάνει με τα προβλήματα, τα πραγματικά των Αιγυπτίων, αλλά για προτάσεις, για παράδειγμα, μείωση του ορίου ηλικία για το γάμο για τις γυναίκες, ή για άλλα θέματα για τα οποία εκφράσαμε ε, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για παράδειγμα, και προσαρμογή κάποιων κανόνων ε, και για τον έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκφράσαμε την ανησυχία μας. Όπως και να έχει, έχουμε εκφράσει ανησυχίες για τα θέματα αυτά και οι Αιγύπτιοι αναρωτιούνται για το τι αποτελεί προτεραιότητα και τι όχι. και χάνουν κάποια από τη δημοτικότητά τους ε, αυτά τα άπειρα μέλη των σαλαφιστών. Με την αντιπροσωπεία μας, λοιπόν, ε, υπό δύσκολες συνθήκες ε, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Ο κύριος Αλσαντάτ ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής, με τον κύριο Σάου, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Μέσων Ενημέρωσης, τον πρόεδρο της ε, δεύτερης, της Κάτω Βουλής. Συναντηθήκαμε, δυστυχώς δεν συναντηθήκαμε με τον κύριο Κατάρτνικ, με τον πρόεδρο της Βουλής, ε, ακριβώς λόγω των, α, της αναστάτωσης που επικρατούσε. Με τον Άλτα Μούσα όμως καταφέραμε να συναντηθούμε με ένα από τα μεγάλα ονόματα από τους υποψηφίους ε, για την ε, Προεδρία. Συναντηθήκαμε που ε, προβάλλεται ως ε, ενδιάμεσος μεταξύ του παλαιού καθεστώτος και της επανάστασης με τους στρατιωτικούς διοργανώσαμε 400 ε, στρογγυλές τράπεζες ε, με γυναίκες εκπροσώπους για ε, των νέων, κόπτες, εκπροσώπους σκεφτικών μειονοτήτων, του επιχειρηματικού κόσμου και διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια των επαφών μας ότι υπάρχει προθυμία για διορθωτικό διάλογο με το Κοινοβούλιο μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε πιο έντονα στην ε, κοινοβουλευτική συνάντηση ε, της Μεσογείου. Ο κύριος Κατάτνικ θα ε, προσκληθεί στις Βρεξέλλες σύντομα και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων έλαβε μία πρόσκληση από τον Έλμαρ Μπρόκ για να έλθει στις Βρυξέλλες. Αναμένουμε λοιπόν ότι θα τον δούμε και στις Βρυξέλλες. Από οικονομικής άποψης, επειδή το θέσατε το ερώτημα αυτό ρητά, η οικονομική κατάσταση δεν είναι τόσο ε, εκθαμβωτική. Ο τουρισμός έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα το τελευταίο έτος. Λιγότερο στη ζώνη την παραθαλάσσια, όπου οι τουρίστες είναι ίσως οι τουρίστες με τα λιγότερα εισοδήματα και εξοδεύουν και λιγότερα στο Κάιρο και στην περιοχή έχει ε, υποστεί δραματική μείωση ο τουρισμός σε ύψος 15% ίσως του συνολικού, ποσοστού, του όγκου. Ε, αναμένεται λοιπόν με ίσως κάποια βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο, παρά τη μείωση του δραματική του τουρισμού, έχει σημειωθεί κάποια οικονομική ανάπτυξη στην Αίγυπτο. Αυτό είναι πολύ θετικό και αυτό σημαίνει ότι η Αίγυπτος μπορεί να σημειώσει σύντομα έντονους ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, σε αυτά θα περιοριστώ και είμαι έτοιμος να ακούσω και τα ερωτήματα των συναδέλφων για να συμπληρώσω αν θέλετε ενδεχομένω ε, στοιχεία. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερ είναι πρώτος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σάιντε Ελκαντράου και να το ρωτήσω αν ε, έπαιξαν ε, τα εξή ρόλο στην επίσκεψή του στην ε, Αίγυπτο. Ξέρετε, συνάδελφε Ελκαντράουι, κατά πάσα πιθανότητα, ότι η Διεθνής Οργάνωση όπως το Ίδρυμα των πολιτιών, Πολιτειών International Republican Institute, το Democratic National Institute, αλλά και αντιστοιχέ οργανώσεις από την Ευρώπη, το Ίδρυμα Conrad Adenauer, που είμαι πρόεδρος ε, στη Γερμανία, αναγκάστηκαν να αναστείλουν ουσιαστικά τις δραστηριότητές τους και το προσωπικό ε, έχει κατηγορηθεί και δύο μέλη του Ιδρύματος Κόνραντ Άντεναουερ ε, έχουν προσαχθεί στο δικαστήριο. Αυτό επηρέασε την επισκεψή σας για τις ιστορικές ε, εξελίξεις ε, στην Αίγυπτο. Είναι σκόπιμο οι επαφές με την Ευρώπη, με την Ευρώπη και με το διεθνές προσκήνιο να συνεχιστούν και θα σας παρακαλούσα να το θέσετε αυτό και σε διαφάρτητα την προσωπία στο Μασρέκ, γιατί αυτό ε, παρεμποδίζει την δημοκρατική εξέλιξη στις χώρες αυτές και η Ευρώπη έχει ρόλο κλειδί. Θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια λοιπόν για την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω Πρόεδρος τον κύριο Πέτερινγκ. Κύριος Μπρέπελς. Κυρία Μπρέπελς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμμετείχα στην αντιπροσωπεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ελκαντράουι για την πλήρη ε, παρουσίαση που μας έκανε. Θα ήθελα, αν μου το επιτρέπει, να προσθέσω κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ε, ανέφερε, αν δεν κάνω λάθος, ε, το γεγονός ότι συνδεθήκαμε με το Γενικό Γραμματέα της Αραβικής Λίγας, ε, του Αραβικού Συνδέσμου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσαμε όχι μόνο για τη Συρία, αλλά και για το ρόλο της Αιγύπτου και του Αραβικού Συνδέσμου στην ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή. Είπαμε σαφήνεια ότι ζήτησε την ε, τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά τον ρόλο του κουαρτέτου, όταν το ρωτήσαμε, δήλωσε ξεκάθαρα ότι θεωρεί ότι το κουαρτέτο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί και θα πρέπει όλα τα καθήκοντα να ε, περάσουν στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας και με τον τρόπο αυτό η δήλωση στη Βεριτό του Αραβικού Συνδέσμου, την οποία δεν σεβάστηκε το Ισραήλ, να μπορέσει να αναπτυχθεί. Ένα δεύτερο σημείο. Ο Σαΐτ μίλησε για μια σειρά προσκλήσεων του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω το εξή ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε ο ίδιος να προσκληθεί και ζήτησα από την Μπάρμπαρα Λόχμπιλερ, από την δική μας πρόεδρος, πρόεδρο, κατά πόσον είναι δυνατόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τις άλλες ομάδες, γιατί έχει καταρτήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης στην Επιτροπή του για το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στο ζήτημα αυτό. Και τέλος, να πω δύο λόγια για τις επαφές μας με εκπροσώπους ε, οργανώσεων γυναικών και νέων, που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Και διαπιστώνουμε ότι είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι για τη σημερινή κατάσταση, γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν ε, υπάρξει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τα οποία πάλεψαν, αγωνίστηκαν στην Επανάσταση και ότι η κυβέρνηση δεν ε, αντιμετωπίζει τα προβλήματα του κόσμου. Εδώ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει φυσικά και το κοινοβούλιο σε μια σύγκρουση. Αυτό ενδεχομένως θα λυθεί αν σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Και τέλο, αν και δεν το είπαμε ξεκάθαρα στα ανακοινωθέντα τύπου, αλλά θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσουμε ανεξάρτητες έρευνες για την ε, βίαιη καταστολή διαδηλώσεων της, ε, από το στρατό. Το ίδιο ζήτησαν και οι Ηνωμένε Πολιτείε και νομίζω ότι θα πρέπει ξεκάθαρα και ρητά να ζητήσουμε διεξαγωγή ερευνών. Και κατά τα άλλα συμφωνώ με αυτά που μας ανέφερε ο Σαΐτ για την αντιπροσωπεία αυτή. La parola alla collega De Η κυρία De Εγώ θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τον Σαΐντ και όλη την αντιπροσωπεία για το ταξίδι που κάνανε και για την παρουσίαση που μας κάνει σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο για μας που δεν είμαστε εκεί και ακόμη όταν είμαστε εκεί να μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα τι γίνεται σε αυτήν την Αιγυπτιακή μεταπολίτευση με στοιχεία ενδιαφέροντα πολλές φορές ή άλλες φορές τρομακτικά. Εγώ δεν άκουσα, δεν κατάλαβα από το Σαΐντ ε, ποιοι παραμένουν ως υποψήφοι για, τους, ε, για, για, πρό, ε, για, για πρόεδρος. Οι σαλαφιστές ε, βγήκαν από τη λίστα, τους γάλανε και εγώ είπα ουφ. Ρωτώ λοιπόν, γιατί για το στρατό και για το πώς ελέγχει τη μεταπολίτευση ο στρατός έχουμε ερωτήσεις. Αν αποκλειστεί ο δικός τους υποψήφιος, ποιον υποστηρίζουν, τι θα μείνει ως υποψήφιος και τι θα κάνει ο στρατός. Είναι αρκετά σημαντικό για μένα. Και εγώ να προσθέσω μία ερώτηση. Καταλαβαίνετε Ιταλικά. Όχι, όχι ακόμα. Σύντομη ερώτηση λοιπόν. Για ποιους λόγους αποκλείστηκε ο, υπο, ο υποψήφιος ε, από την προεδρική κούρσα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο. Αν σωστά έχω καταλάβει, δέκα είναι υποψήφια για την προεδρική θέση. Από διαφορετικά προσκήνια και τρεις ε, είναι, αν θέλετε, τα φαβορή. Φουτού, που υποστηρίζεται από τους αλαφιστές. που θεωρείται μετριοπαθής μουσουλμάνος και υποστηρίζεται και από τους bloggers. Μπορεί να ενσωματώσει την ανανέωση, αν θέλετε, του συστήματος από πλευράς κυβερνητικής και στρατιωτικής, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ε, ο οποίος ε, είναι υποψήφιος και έχουμε και τον υποψήφιο της αδελφότητας των μουσαλμάνων, και ο μία από τις λίγες ε, φιγούρες που είναι γνωστός ε, εκτός Αιγύπτου και σε όλη την Αιγύπτο. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά τίποτα, αλλά στις δημοσκοπήσεις ε, σημειώνει πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτοί οι τρεις-τέσσερις λοιπόν υποψήφοι, τέσσερις υποψήφοι είναι αυτοί που ξεχωρίζουν. Έχουν εξαιρεθεί όντω κάμποσα άτομα και ο υποψήφιος των σαλαφιστών έχει αποκλειστεί επειδή η μητέρα του έχει διπλή υπηκότητα. Είναι Αιγύπτια και Αμερικάνα. Αυτό αποτελεί λόγο αποκλεισμού για την Επιτροπή την Εκλογική. Είναι μάλλον τυπικό το ζήτημα και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Αυτό ψάξανε και βρήκανε ένα λόγο να το αποκλείσουν. Γίνονται λοιπόν ελιγμοί. Αυτός είναι όμως ο επίσημος τυπικός λόγος για τον οποίο ε, αποκλείστηκε. Γιατί έχει θεσμούς μέσω της μητέρας του με, του, με τη ΣΥΠΑ. Για να επανέλθω σε αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος Πότερινγκ. Να σας επιβεβαιώσω ότι σε ζητήματα μη κυβερνητικών οργανώσεων και ε, ιδρυμάτων ε, ήταν πολύ προβεβλημένα τα θέματα αυτά στις συζητήσεις μας. Το τονίσαμε και ζητήσαμε εξηγήσει σε πολλές περιπτώσεις και στο ε, ανακοινωθέν τύπου τα αναφέραμε αυτά. 25 δημοσιογράφοι παρευρέθηκαν πολλοί δηλαδή, ήταν καλή προσέλευση των δημοσιογράφων. Γιατί λοιπόν προκλήθηκε αυτή η κατάσταση. Θεωρούμε ότι το στρατιωτικό καθεστώς ήθελε να κερδίσει δημοτικότητα εις βάρος τέτοιων ιδρυμάτων, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι είμαστε κατά της αλλοδαπής παρέμβασης ε, από όπου και αν προέρχεται από ιδρύματα, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το χάος που επικρατεί για να υποστηρίξουν κάποιες, ε, κάποια πολιτικά κόμματα κτλ. Και αυτό είχε αντίκτυπο στην Αίγυπτο. Και υπό τη μορφή υποστηρίξης μας λένε. Αλλά φυσικά έχει προκύψει και πάρα πολύ κριτική. Και διαπιστώνει ο κόσμος ότι παραπήγε αυτή η κατάσταση. Συζητιέται αυτή τη στιγμή ένα καινούργιο νομοσχέδιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στο Κοινοβούλιο που ψάχνει τρόπους επίλυσης των θεμάτων αυτών. Θα τεθούν και κάποιοι όροι για την διαφάνεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ούτω καθεξής και σε ό,τι αφορά χρηματοοικονομική διαφάνεια. Κανείς όμως δεν πρόκειται να εξαιρεθεί στο μέλλον. Εμείς συνομιλήσαμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με ανθρωπιστικές οργανώσεις σε ό,τι αφορά το πνεύμα του νέου νομοσχεδίου και μας αναφέρουν ότι η στιγμή δεν είναι καλή για να συζητηθούν τέτοια ζητήματα, γιατί βρισκόμαστε τρεις εβδομάδε από τις προεδρικές εκλογές και ο σημερινός ε, νόμος για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις παρέχει ένα σωστό πλαίσιο λειτουργίας, δεν υπάρχει κάποιος λόγος προσαρμογής, εκτός κι αν ε, προηγηθεί μία ε, περίοδος περισυλλογής, σωστή. Ο σχετικός νόμος που ισχύει στη Λιβύη θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ θετικός. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου κάποιες δυνάμεις θέλουν να εκμεταλλευτούν από ό,τι φαίνεται την κατάσταση, την περίσταση, για να δυσκολέψουν το έργο κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Και θέλουν να ενισχύσουν την, ε, τον έλεγχο των αρχών στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η κατάσταση, αλλά από ό,τι μας είπε ο Ελ Σαντάτ, ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ότι τα πράγματα θα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα άτομο λογικό, ο οποίος όντως θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να μεταβεί στις Βρυξέλλες, να μας επισκεφτεί. Αλλά φυσικά δεν είδαμε κανένα κείμενο και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που έχει ανοιχτό τέλος. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Το θέσαμε όμως το ερώτημα και το παρακολουθούμε δελεχώς. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και για τις απαντήσεις. Τώρα παρουσίαση του Έμερ Κοστέλο για την Παλαιστίνη και από τη, συνεδρίαση που είχα, από τη συνάντηση που είχαν με, την, με το νομοθετικό Παλαιστινιακό Συμβούλιο από τις 2 ως 5 Απριλίου. Τώρα ο κύριος Κοστέλο για λόγους ε, εργασίας δεν είναι παρόν. Θα το παρουσιάσει η κυρία Αουκέν που είναι αντιπρόεδρος αντιπροσωπείας. Λέγαμε, είπαμε ότι επισκέφθηκαν σε αυτές τις ημερομηνίες την Ιερουσαλήμ και τα κατεχόμενα. Παρακαλώ λοιπόν να μας ε, κάνετε την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και βέβαια ο κύριος Κοστέλο δεν μπορούσε να είναι παρόν. Σας ζητά συγγνώμη. Πέντε μέλη της αντιπροσωπείας μας ήταν από διαφορετικές χώρες, από Πέντε χώρες και τέσσερα κόμματα. Ένα από τα μέλη μας ήταν μέλος και της αντιπροσωπείας του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Και όταν είδε τι έγινε ε, και το αναφέραμε στην δήλωσή μας στον τύπο. Είναι πάρα πολύ σύντομη η δήλωσή μας, περιλαμβάνει όλα τα συμπεράσματα αυτά και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πολύ καλή αποστολή. Και πάρα πολύ εύστοχη. Πρέπει να πω όμως ότι, συγγνώμη που σας τα λέω αυτά, αλλά η κοινική στρατηγική της Ισραηλινής κυβέρνησης φαίνεται να επιτυγχάνει. Στο Ισραήλ τουλάχιστον. Η Παλαιστίνη δεν υπάρχει πια. Η Παλαιστίνη <clears throat> είναι διχασμένη σε 4-5 κομμάτια πια, δεν είναι ενιαίο έδαφο. δεν υπάρχει καμία εδαφική συνοχή και ενώ υπάρχουν οι περιοχέ α, β και γ από τις συμφωνίες του Όσλο, που αυτό υποθέτει να ήταν μια ενδιάμεση διαρρύθμιση, η περιοχή Γ είναι περιοχή που θα προσαρτηθεί, προσαρτηθεί από το Ισραήλ, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να παρισφρεί και στις περιοχές Α και Β υποσκάπτοντας την εξουσία των Παλαιστινίων. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να διατηρήσουμε την εντύπωση ότι θα μπορούσε να προκύψει μια λύση δύο κρατών που θα ζουν δίπλα-δίπλα μέσα σε συνθήκες ειρήνης, σε αναγνωρισμένα σύνορα, όπως υποτίθεται ότι θέλουμε. Και θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα ότι και τα λεφτά των ε, φορολογούμενών μας απλώς δημιουργούν υποδομές για τους Παλαιστινίους που με μεγάλη χαρά μετά καταστρέφουν οι Ισραηλινοί και δεν μας δίνει κανείς πίσω τα λεφτά μας. Η Γερμανία, η Δανία, η Πολωνία θα έπρεπε κάποια στιγμή να ζητήσουν πίσω τα χρήματά τους όταν το Ισραήλ καταστρέφει τις υποδομές που έχουμε δημιουργήσει. Νομίζω ότι η αντιπροσωπεία μας εξακολουθεί να υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών. όχι μόνο για το καλό της Παλαιστίνης αλλά και για το καλό του Ισραήλ. Γιατί κανείς δεν βλέπει να υπάρχει προοπτική ούτε για την Παλαιστίνη ούτε για το Ισραήλ αν δεν υπάρξει μια λύση. Δηλαδή υπάρχουν προοπτικές για το μέλλον αλλά δεν είναι ευίωνες. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ πιο στεναροί. Δεν το θέσαμε έτσι στο κείμενο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Όσλο πέθανε. Δεν λειτουργεί. Και τώρα χρησιμοποιείται μονάχα σαν πρόσχημα για την κατάσταση που επικρατεί. Επίσης αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι ότι κοιτάξαμε και το θέμα των κρατουμένων. Είχαμε αντιμετωπίσει το θέμα αυτό προηγουμένως και παρακολουθούμε τον πολίτη αυτό της Δανίας, ο οποίος είναι εκεί κρατούμενος σε απεργία πίνης και λέμε πόσο αρνητική είναι η κατάσταση. Μα είναι πάρα πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε υποδικητική κράτηση, εκατοντάδε και γι' αυτό το λόγο κάνουν απεργία πείνα. Κάποιοι από αυτού πεθαίνουν. Τι θα αρχίσει να είναι κοντά στο θάνατο, τι θα γίνει αν πεθαίνουν και παρόλα αυτά το ανώτατο δικαστήριο της, του Ισραήλ δεν αντιμετωπίζει τις περιστάσεις, τις περιπτώσεις τους. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν του, του πληθυσμού της Παλαιστίνης είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Πρέπει όμως να κάνουμε κάτι και να το κάνουμε γρήγορα και με τρόπο στεναρό. Υπάρχουν τα 203 παιδιά τα οποία είναι στη φυλακή. Για να καταλάβετε τι γίνεται, αλλά το ξέρετε ήδη πολλοί από εσά. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τη συνάντηση με το κουαρτέτο, με την τετραμερή σύνοδο και εδώ είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη δύναμη στο κουαρτέτο που είναι πρόθυμη να κάνει κάτι. Έχουμε κάποιες συστάσεις εδώ και μπορώ να σας τις αναφέρω. Χωρίς να υπάρξουν εμπάργο και κυρώσεις και όλα αυτά, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εφαρμόσει την νομοθεσία για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί από επίκους να μην μπορούν να την χάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης, γιατί αυτό είναι καταρχήν παράνομο. Εναπόκειται στο Ισραήλ να το εξασφαλίσει αυτό ότι συμβαίνει, αλλά δεν εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Είναι θέμα της Κομισιόν να πει στο Ισραήλ δεν είναι θέμα μονάχα τοθεσίε, αλλά ότι πρέπει να εξασφαλίσει ότι κανένα προϊόν από τις κατεχόμενες, τα κατεχόμενα εδάφη δεν την χάνει προτιμησιακή μεταχείριση. Επίση πρέπει να κάνουμε σαφέ ότι αν αναβαθμίσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με το Ισραήλ, θα στείλουμε ένα πολύ αρνητικό μήνυμα στην Παλαιστίνη. Θα δουν ότι ανταμείβουμε το Ισραήλ. είδαμε ότι το Ισραήλ ζητάει όλο και περισσότερο, ότι ζητάει περισσότερα, αλλά τώρα παίρνει περισσότερα χωρίς να έχει δώσει τίποτα. Αν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, θα δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραγνωρίσει, έχει ξεχάσει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Επίσης θα πρέπει να θεωρήσουμε το Ισραήλ οικονομικά υπεύθυνο όταν καταστρέφονται τα προϊόντα μας. Να πούμε ότι θέλουμε τα λεφτά μας πίσω. Πρέπει όμως να πούμε στα κράτη-μέλη μας ότι δεν έχουμε μια κοινή πολιτική. Και το ξέρετε αυτό. Πολλές φορές όμως δρούμε σαν να υπάρχει μια τέτοια κοινή πολιτική και απλώς αφήνουμε δύο-τρία κράτη μέλη να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω τη συνάντηση που είχαμε με τον δικό μας πρεσβευτή, ο οποίος μας είπε ότι οι Παλαιστινοί δεν χρησιμοποίησαν την ευκαιρία που είχαν στην ε, Γενική Συνέλευση και θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει αν δεχόντουσαν αυτή την προσφορά ότι θα τους υποστηρίξουν τα άλλα κρατημέλη. Μα ήταν μια κενή πρόταση αυτή. Και δεν μπορούσε ο Μαχμού να γυρίσει πίσω στο λαό του και να πει ότι θα υπήρχε μια υποστήριξη η οποία δεν σήμαινε τίποτα. Μια αναβάθμιση θα πρέπει να τους ευθυγραμμίσει τουλάχιστον με το Βατικανό. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από όλα τα κρατημέλη να συνενέσουν σε κάτι τέτοιο, γιατί στο στον ΟΗΕ λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε επίπεδο κρατών, εθνικών κρατών. Και καταλαβαίνουν οι Παλαιστίνοι ότι όταν χρησιμοποιούν βία, τους καταδικάζουν. Αν χρησιμοποιούν ειρηνικά μέσα, τους αγνοούν. Τους καταδικάσαν γιατί πήγαν και στον ΟΗΕ με ειρηνικά βήματα για να πετύχουν κάτι. Ακολουθήσανε όλους τους κανόνες. Και αντί να τους επενέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους τιμωρεί. Και πρέπει να τους πούμε χρησιμοποιήστε το διεθνές πλαίσιο. Και επίσης θέλω να σας αναφέρω κάτι το οποίο το γνωρίζετε ήδη. Το Δεκέμβριο 2009 όλοι οι υπουργοί εξωτερικών μας είχαν κάνει μια ομόφωνη δήλωση η οποία ήταν πολύ καλή και αξίζει να τη διαβάσετε από όλου του υπουργού μα. Και ίσως πρέπει να την πάρουμε σοβαρά αυτή τη δήλωση. Οπότε ας δεχτούμε και ας ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι έχουμε και <clears throat> τέσσερις εκθέσεις που έχουν δημοσιευτεί σε σχέση με τους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ. Και η καλύτερη ήταν αυτή που αφορούσε την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Υπήρχαν πολλές καλές συστάσεις λοιπόν στα κράτη-μέλη. Είχαμε μια σύσταση για την περιοχή Γάμα του Όστο. Και αυτό το οποίο λέμε τώρα ήταν πολύ κοντά στην προηγούμενη έκθεσή μας. Και επίσης για τη βία που ασκείται από τους επίκους. Γιατί οι έπικοι είναι σκοτώνουν, δεν καταστρέφουν μονάχα ιδιοκτησίες, δεν ξεριζώνουν ελιές, αλλά σκοτώνουν κιόλας, είναι ένοπλοι. Κανείς δεν θεωρεί ότι είναι τρομοκράτες, ούτε καν ε, αγωνιστές για κάποιο στόχο, αλλά είναι ένοπλοι και πυροβολούν και σκοτώνουν. <clears throat> Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναφέρει τα ονόματα αυτών των βιαίων επίκων και να πούμε ότι δεν τους δεχόμαστε στις χώρες μας. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο λοιπόν αν είχαμε τουλάχιστον ένα κατάλογο αυτών των επίκων. Αν δεν δράσει όμως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον να ξεχάσετε αυτό το όραμα των δύο κρατών. Τα πράγματα είναι ειρηνικά στην Παλαιστίνη. Εδώ για πολύ καιρό, πολύ λίγα επεισόδια σε σχέση με αυτά τα οποία υφίστανται. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχουμε τόσα επει, επεισόδια. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα και δεν τους δώσουμε κάποια ελπίδα, <clears throat> τι θα γίνει όταν υπάρχει μια πραγματικά μια επίθεση σε ειρηνικέ διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ, τι θα γίνει στην Αίγυπτο. Τι θα γίνει στον αραβικό κόσμο δεν θα είναι μοναχα διαδηλώσεις, αλλά τα πράγματα θα γίνουν πολύ σκληρότερα. Αυτά τα οποία βλέπουμε τους τελευταίους μήνες είναι σαν το προήμιο μιας νέας συντηφάδα. Είναι σαν και αυτά τα οποία είδαμε πριν από τη δεύτερη εντιφάδα. Πρέπει να κάνουμε κάτι λοιπόν πολύ γρήγορα. Πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι να δείξει ανησυχία η ε, συντριβή ή οτιδήποτε τέτοιο, όταν το Ισραήλ εξακολουθεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και σας προτείνω να διαβάσετε το, την έκθεσή μας και σας παρακαλώ μην προχωρήσετε στην αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ. Θα στείλει ένα πολύ κακό μήνυμα σε όλη την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Μάργαρετ Όκεν μιλάει σε μια αίθουσα που είναι λίγο άδεια σήμερα. Έθεσε ένα θέμα το οποίο εμένα με, με, με, με ταλαιπωρεί. Για τη βία τη βία των επίκων που έχει καταγραφεί και από οργανώσεις του ΟΗΕ και μου θύμισε και έναν Παλαιστίνιο φοιτητή που έκανε που κάνει το δοκτορά του στις πολιτικές επιστήμες και ήρθε να μου κάνει μία ερώτηση στο γραφείο μου που με δυσκολία μπορούσα να απαντήσω. Οι συνάδελφοί σας, οι βουλευτές σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εκτιμούν το γεγονός ότι οι δικές μας ε, διαδηλώσεις είναι μη Δηλαδή, εσείς υποστηρίζετε τη μη βία. Φυσικά και Και, αυτή η ερώτηση με, με, με δυσκόλεψε. Γιατί φυσικά είμαστε εμείς κατά της βίας. Και θεωρώ ότι σήμερα όπως έχει κατάσταση στην Παλαιστίνη η στάση των Παλαιστινίων είναι μία στάση μη βίας. Ε, όταν η Μάργαρετ μιλάει για ένα μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε, πρέπει κάπου να, κάτι να κάνουμε ούτως ώστε να παραμείνει αυτό το, το, το, το στοιχείο της μη βίας. Αυτή η νέα γενιά που βγαίνει είτε είναι από τη Φατάχ, είτε από τη Γάζα, είτε από την Χαμάς, δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να λέμε εμείς ότι είμαστε κατά της βίας, χωρίς, ε, άμα εμείς δεν τους στείλουμε και ένα μήνυμα σαφές, για αυτή την επιλογή. Άμα δεν του στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, κινδυνεύουμε να μην μας καταλάβουν καθόλου. Μάργαρετ, επανέρχομαι σε αυτό. Δηλαδή, να, αυτός ο φοιτητή μου έλεγε, Μα καταλαβαίνετε τι γίνεται. και μέχρι πού θα καταφέρουμε εμείς να συνεχίζουμε να έχουμε μία ειρηνική ύπαρξη. Ο Πρόεδρος Πέτερινγκ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Μάρκρετ Άουκεν για την παρουσίαση αυτή που μας έκανε και την έκθεσή της ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πάντα ε, εκπροσωπούμε την άποψη ότι το Ισραήλ θα πρέπει να έχει ασφαλή σύνορα και το ίδιο και για, θα πρέπει να ισχύει και για την Παλαιστίνη. Δύο κράτη λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα πρέπει να έχουν την αξία τους, την ανθρώπινη αξία τους, αλλά την ίδια ανθρώπινη αξία έχουν και οι Παλαιστίνοι. Και σήμερα τη βλέπουμε με την ε, επέκταση των επικισμών. Η βάση για ένα Παλαιστινιακό κράτος ε, καταστρέφεται ουσιαστικά. Και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μεγάλο διακύβευμα και είναι νομίζω προς το συμφέρον και του ίδιου του Ισραήλ, γιατί όλο και πιο πολύ διαβάζουμε ότι είναι οι Παλαιστίνοι σήμερα βγαίνουν και λένε ότι αν έχουμε ένα κοινό κράτος, οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί, κάποια στιγμή οι Παλαιστίνοι θα σχηματίσουν την πλειοψηφία γιατί έτσι είναι τα δημογραφικά στοιχεία. Μετά από συνάντηση με Παλαιστίνιους, ακούμε ότι αν δεν πραγματοποιηθεί η λύση του διπλού κράτους και σχηματιστεί ένα κράτος με το Ισραήλ, θα βρεθεί σε μια κατάσταση το Ισραήλ, σε μια δύσκολη κατάσταση, όπου θα, τι θα κάνει, θα δημιουργήσει ένα apartheid όπως στην Νότια Αφρική. Αυτό ως πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα αν υπάρξει κράτος στην Παλαιστίνη, χρειάζεται και ειρήνη και κατανόηση μεταξύ Φατάχ και Χαμάς. Ποια ήταν λοιπόν η εντύπωση της αντιπροσωπείας σε ό,τι αφορά τη σχέση αυτή Φατάχ και Χαμάς. Κανένας άλλος δεν θέλει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους Είναι πράγματι σκάνδαλο το ότι δεν αναγνωρίζουμε περισσότερο τις ειρηνικέ ε, διαδηλώσεις και δεχόμαστε να τις αντιμετωπίζουν με δακρυγόνα, με κρατήσεις κτλ. Και εγώ ήμουνα στη Βιθλέμ πέρσι και τα είδα αυτά και δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. Και φυσικά με αντιμετωπίσαν πολύ καλύτερα από τους άλλους διαδηλωτές. Αλλά η προσπάθεια που έγινε στον ΟΗΕ ήταν μια ειρηνική κίνηση και δεν είναι σωστό να τους αντιμετωπίσουμε σαν να είναι τα κακά παιδιά. Όλη αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τους αποστερεί από κάθε ευθύνη, από κάθε ελπίδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτά τα ελληνικά μέσα. Θέλω να προσθέσω εδώ αυτό που είπε ο Hans για τις προοπτικές που ανοίγονται. Αυτό το οποίο λένε τώρα είναι ότι ο Νετανιάχου τώρα χρησιμοποίησε τον όρο δύο κράτη. Υποστηρίζει τα δύο κράτη. Τα δύο κράτη όπως είναι τώρα βέβαια. Μα έχουμε αυτή τη στιγμή το μισό πληθυσμό να ζει σε απόλυτη ευμάρεια, και να, κατα... να καλλιεργεί τη γη του κτλ. Και οι άλλοι να είναι περιορισμένοι σε όλο και μικρότερα θυλάκου που δεν έχουν επικοινωνία. Δεν υπάρχουν καμία ελπίδα για το μέλλον. Και όταν μιλάμε με τους Ισραηλινούς βλέπουμε ότι φοβούνται και αυτοί όπως και εμείς για το μέλλον. Από την άλλη πλευρά μας από τους Παλαιστινίους ούτε καν συζητάνε για το μέλλον. Είναι, καν, είναι σαν να μην υπάρχει καν στο παιχνίδι το τι θα γίνει στο μέλλον. Ελπίζω ότι η Ευρώπη και ο υπόλοιπο κόσμο δεν θα δεχτούν αυτά τα πράγματα. Το ελπίζω πραγματικά. Θα μπορούσε να προκύψει ένα μοντέρνο και κοσμικό κράτος το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχετε τόση ματέωση που νιώθει ο, πολιτισμό, ο Έχετε τους νέους οι οποίοι έχουν δει φαντάρους του Ισραηλινού στρατού να σκοτώνουν τους γονείς τους. Είναι οι μόνες εικόνες που έχουν από το Ισραήλ. Αν αυτό δεν είναι συνταγή για τρομοκρατία, τι είναι. Είναι εντυπωσιακό που δεν έχουμε περισσότερη τρομοκρατία. Όταν συζητάτε με τους ε, ιερωμένους στην Παλαιστίνη, τους επικεφαλείς των θρησκευτικών ομάδων, ναι, προσπαθούν πράγματι να εκπαιδεύσουν τη νέα γενιά, να έχει κάποιες αξίες, να έχει πνευματικότητα, να βλέπουν το μέλλον καλύτερα και είναι τεράστιο το έργο που γίνεται από αυτές τις ομάδες τις θρησκευτικέ στην Παλαιστίνη, αλλά δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχουν προοπτικές αν δεν κάνουμε κάτι. Το Ισραήλ δεν ασχολείται καθόλου με το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Αναφερθήκατε στην συμφιλίωση, μιλήσαμε για τη συμφιλίωση Φατάχ και Χαμάς. Δυστυχώς το Κοινοβούλιο όμως ποτέ δεν δέχτηκε την ιδέα του ότι δεν πρέπει να μιλάμε τη Χαμάς ή ότι δεν έπρεπε να αναγνωρίσουμε την εκλογική νίκη της Χαμάς. Αλλά κάθε φορά που γίνονται προσπάθειες για συμφιλίωση μεταξύ των δύο πλευρών της Φατά και της Χαμάς, τους τιμωρούν. Λέει το Ισραήλ, α, δεν θα ξαναμιλήσω μαζί σας. Και αυτό το δεχόμαστε. Εκεί που έχουμε ζητήσει αυτή τη συμφιλίωση εμείς, δεχόμαστε αυτή την αντιμετώπιση του Ισραήλ. Αφού έχουμε πει ότι η Αίγυπτος και η Ορδανία έχουν κάνει πολύ καλά να βοηθήσουν αυτή τη συμφιλίωση. Προφανώς υπάρχουν ομάδες που δεν θέλουν μια τέτοια προσέγγιση. Η ακραία πτέρυγα της Χαμάς, οι σαλαφιστές όλοι αυτοί δεν θέλουν να υπάρξει συμφιλίωση. Προτιμούν την αντιπαράθεση και από την άλλη πλευρά αντιστοίχως. ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, <clears throat> είπαν ότι «Α, αν συμφιλειωθείτε θα σας κόψουμε τη χρηματοδότηση». Όταν η, έγινε η ψηφοφορία στην UNESCO για την ε, αναβάθμιση της θέσης του, των Παλαιστινίων, κόψαν τη χρηματοδότηση. Το Ισραήλ βέβαια παραμένει στην UNESCO γιατί δεν θέλει να χάσει την δυνατότητα πίεσης του αλλά κοπήκανε όλες οι χρηματοδοτήσεις προς την Παλαιστίνη. Το Ισραήλ κατακρατάει φορολογικά έσοδα. Τι του είπαμε. Όχι, όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Μήπως θα θέλατε, μήπως θα ήσασταν τόσο ευγενικοί να δώσετε πίσω αυτά τα λεφτά εκεί που ανήκουν. Μερικές φορές είμαστε υπερβολικά αυρόφρονες. Πρέπει να κάνουμε κάτι όμως. Αυτό το ξαναλέω. Αυτή είναι η σύστασή μου. Διαβάστε λοιπόν τις τέσσερις εκθέσεις από τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Δεν είναι μακροσκελής, έχουν πάρα πολλά παραδείγματα, ιδίως αυτή από την Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει πολύ καλές συστάσεις για το τι μπορεί να γίνει ειρηνικά, χωρίς να τιμωρήσουμε κανένα. Ειρηνικά για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί υπάρχουν και από την Παλαιστίνη και από το Ισραήλ ακόμα άτομα που είναι προσιλωμένα στην ιδέα των δύο κρατών αλλά δεν, μάλλον για ένα κράτος, για ένα ενίο κράτος, δεν είναι όμως ρεαλιστικά αυτά τα πράγματα. Γιατί ήδη τώρα έχουμε ουσιαστικά ένα κράτος. Γιατί λοιπόν δεν προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα στην Παλαιστίνη πραγματικά για τους νέους είναι τραγικά. Και ακόμα και αυτοί από τους, ε, τις θρησκευτικέ οργανώσεις έχουν εντυπωσιαστεί από το πόση ελπίδα ξεκολουθεί να υπάρχει. Και να απαντήσω στη Βερονίκα όταν μίλησε για την αντιμετώπιση που δεν είναι βία. Παλιά ο ηρωάς μας ήταν ο Νέλσον Μαντέρα. Γιατί δεν βγήκε από τη φυλακή τότε. Γιατί δεν ήθελε να απαρνηθεί τη βία. Γι' αυτό έμεινε στο Ρόμπιν Άιλαντ στη φυλακή τόσο καιρό, γιατί δεν έχει απαρνηθεί τη βία. Και οι Παλαιστίνοι έχουν απαρνηθεί τη βία και τελικά ανταμείβει αυτό το Ισραήλ. Κάτι όμως μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο. No, al punto. Δεν πάμε στο επόμενο σημείο. Γιατί λείπει ο Νίκολας Βέσκοτ. Ε, Διάλειμμα. Δεν έχουμε νέα του κυρίου Βέσκοτ. Δεν καταφέρνουμε να τον βρούμε. Και δεν μπορούμε να προβλέψουμε και πόσες ώρες θα αργήσει ο κύριος Βέσκοτ. Η συνάδελφος Δεκάιζερ ζήτησε το λόγο για δύο λεπτά Και αν συμφωνείτε να την ακούσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για να εξηγήσω τι ήθελα να ζητήσω από τον αντιπρόσωπό μας. Εδώ και ένα χρόνο μετά από την ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν για την οποία εργαστήκαμε αγρίως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, βάλαμε λεφτά, βάλαμε τεχνική βοήθεια. Υπήρξε μια τεράστια διακριτικότητα, για να μην πω τίποτα άλλο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή τη χώρα. Γνωρίζουμε, η κυρία Άστον, υποστήριξε το πάνελ υψηλού επίπεδου του ΕΛΜΠΕΚΙ της Αφρικανικής Ένωσης. Αλλά δεν κατέληξαν ποτέ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βορρά και Νότου και η κατάσταση τελικά έχει εξελιχθεί σε μια κατάσταση ε, ιδιαίτερα εκρηκτική, προπολεμική κατάσταση θα λέγαμε. Πέρα από μερικά σκόρπια ανακοινοθέντα της ε, κάτι άστον και μετά την, το ανακοινοθέν του ΟΗΕ που και η κάτι άστον μετά έκανε, μία, μία, έκανε μετά μια άλλη δήλωση δεν βρίσκω πουθενά αλλού οποιοδήποτε χνάρι. Έχει χαθεί η ορατότητα. Βλέπουμε τους Κινέζους που βάλανε 8 δις δολάρια στο τραπέζι για μια άλλη pipeline και παρενέβησαν μαζικά γιατί ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο. Αυτή η κατάσταση, η εμπόλεμη κατάσταση με μια δραματική ανθρωπιστική κατάσταση συνδεδεμένη με το πρόβλημα του πετρελαίου. Θέλω να ξέρω ποιες είναι οι επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι εκεί μέσα έχουν κάνει αυτή τη χώρα πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη ορατότητα και περισσότερη ενημέρωση για, για, το που βρισκόμαστε εκεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουμε αποκλειστεί από το όλο παιχνίδι. Και αυτό ήθελα εγώ να αναφέρω στον εκπρόσωπό μας. Και αν δεν είναι δυνατόν, θα ήθελα, εντάξει τώρα είναι πόλεμος, ε, έχουμε ένα νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάπαυση του πυρός, εδώ και μερικές μέρες αρχίζουν και μορφοποιούνται τα πράγματα. Θα ήθελα να θα ήθελα να τεθεί το ερώτημα αυτό για την ανθρωπιστική πολιτική οικονομική σημασία στην επόμενη ολομέλεια και να ζητήσουμε λογαριασμούς και ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Σε πολλές εκθέσεις ε, για τις εκλογές και ο κύριος Αλαφράνκα δεν είναι εδώ. Λέμε πάντοτε ορίστε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη μεταβατική περίοδο, τη μεταπολιτευτική περίοδο μιας χώρας, να την συνοδεύσουμε στην προκειμένη περίπτωση του Σουδάν. Δεν ε, παρακολουθήσαμε αυτή τη μεταπολιτευτική φάση. Βλέπω τον Τσαρστάνο, ο οποίος από πολύ κοντά παρακολούθησε πάντα το θέμα του Σουδάν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλό θα ήταν να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα σε αυτό το ζήτημα και να ζητήσουμε περισσότερες εξηγήσει για το πώς χάθηκε δηλαδή από την επικαιρότητα αυτό το θέμα. Ωραία. Δράτουμε αυτό το αίτημα της κυρίας Δεκάιζερ και θα ενημερώσουμε σχετικά. Τώρα, στις 14 Μαΐου ο ειδικό μας εκπρόσωπος για το Σουδάν, η κυρία Μάρσμπεν θα είναι παρούσα και είναι ευκαιρία για να εκφράσουμε τις γνώμες σας. Ε, ευχαριστώ όλους σας για την υπομονή σας, αλλά επειδή δεν είναι διαθέσιμος ο κύριος Γουέσκοτ, ε, το αναβάλουμε για την επόμενη φορά. Ευχαριστώ.